Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συνάδελφοι. <laughs> Πρώτο θέμα της ημερήσιας διέταξης έχουμε έγκριση. έχετε λάβει όλοι αντίγραφο. Την εγκρίνουμε. Και αν ναι, μπορώ να περάσω στο επόμενο θέμα τη τη διάταξη, που είναι το Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Δίκτυο για Ανταγωνιστικέ Απορρευματικέ Μεταφορέ, με εισηγητή τον κύριο Μαρινέσκου. Είστε εδώ. Τι έχετε διαδικαστικό. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στο φύλλο της γραμματείας δείχνει ότι πρώτα ψηφίζουμε, Πρόεδρε. Όχι ότι συζητούμε την έκθεση Μαρινέσκου. Δεν μου είπε κανείς ότι άλλαξε η μερίσια διάταξη. Και ξέρετε ότι έχουμε και άλλες συνεδριάσεις που συμπίπτουν. Δεν ξέρω γιατί ε, έγινε η αλλαγή, αλλά πάντως εμείς ήρθαμε για να ψηφίσουμε τώρα. Πρώτο θέμα. Πρόεδρος, κύριε Μπράντμπερν, εγώ ξέρω ότι η ψηφοφορία για την ασφαλή της πολιτικής αεροπορίας είναι στις 3 και 4. 3 και 50, συγγνώμη. Αυτό ξέρω ότι συμφώνησε στη τελευταία του συνεδρία οι συντονιστέ. Μπορούν να μου το επιβεβαιώσουν παρακαλώ. Βλέπω ότι οι συνάδελφοι γνέφουν καταφατικά. Άρα να ακούσουμε πρώτα αυτό και μετά να επανέλθουμε για την ψηφοφορία. Κύριος Μπράτμορ. Δεν ξέρω αν άλλαξαν ε, τα χρονοδιαγράμματα. Πάντως ούτε η κυρία Φώστερ ούτε εγώ δεν ενημερωθήκαμε. Και παρακαλώ να ενημερωνόμαστε εγκαίρως. Ε, ναι κύριε Μπράντμπορν, κατανοώ το επιχείρημά σας, έχετε δίκιο σε αυτό. Απλά φαίνεται ότι οι περισσότεροι ε, συνάδελφοι έχουν αντιληφθεί διαφορετικά την ημερήσια διάταξη στην οποία συνεφώνησαν οι συντονιστές. Λυπούμε για την όποια δυσκολία σας προκαλεί αυτή η παρεξήγηση, αλλά αυτή είναι η μερίσια διάταξη. Κύριε Μαρινέσκου, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Πού είστε? Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά με τους ε, διαδρόμους ε, διακίνησης εμπορευμάτων μιλάει για τους όρους και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν για τη δημιουργία ενός τέτοιου σιδηροδρομικού διαδρόμου διακίνησης εμπορευμάτων και των όρων επίσης που η Κομισιόν χρειάζεται για να εγκρίνει τη δημιουργία του. Στην πρόταση λοιπόν του Συμβουλίου θα δημιουργηθούν ορισμένοι διάδρομοι στο βαθμό που θα ξεκινήσει να ισχύει ο, κανονισμός. Έχουμε λοιπόν εννέα διαδρόμους. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά μεταξύ της ερμηνείας που δίνει το Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου. Λοιπόν, η ενία θηρίδα. Κατά τη γνώμη μου αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θέλουν να υπάρχει μία ενιαία θηρίδα όπου οι ε, τούντες μπορούν να ζητούν ένα διάδρομο, ένα πέρασμα για ένα διεθνές τρένο εμπορευμάτων αλλά η θηρίδα, αυτή η ενιαία θηρίδα μπορεί να αντικατασταθεί απόλυτα από τις ήδη υπάρχουσες σιδηροδρομικές υπηρεσίες και η ενιαία θηρίδα μπορεί να λειτουργεί για άλλες υπηρεσίες. Επίσης υπάρχει και ένα πρόβλημα σχετικά με, τις, ε, με το τι εννοούμε εμείς ε, ε, εμπόρευμα προτεραιότητες, ναύλος προτεραιότητες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα, πώς να ορίσουμε εμείς, πώς ε, να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες όταν υπάρχει, μια, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφορίας. Το κοινοβούλιο θέλει τα επιβατικά τρένα να είναι αυτά τα οποία θα έχουν απόλυτα την προτεραιότητα πάντα. Ενώ το Συμβούλιο θέλει να κρίνουμε από τη διάρκεια της καθυστέρησης του δρομολογίου για την επιλογή του τρένου. είτε είναι επιβατικό είτε, είτε μεταφέρει εμπορεύματα. Υπάρχει τώρα και κάτι άλλο. Λοιπόν, θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι η ενία θηρίδα είναι και η προστιθέμενη αξία όλης αυτής της έκθεσης. Τώρα για τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα διαπραγματευτούμε περισσότερο με το Συμβούλιο. Θα συναντηθούμε εμείς με το Συμβούλιο αύριο. Το πρόγραμμα έχει ήδη προταθεί και ελπίζουμε να σεβαστούμε και τις 45 μέρες για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Σε ευχαριστώ κυρία Μαρινέσκου. Η κυρία Μπιλμπάου πρώτα γιατί ο κύριος Αλχαντράουι δεν έχει καθίσει ακόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μαρινέσκου μας έκανε μια πολύ καλή περίληψη για το που έχουμε διαφορές. Εμείς είχαμε μια συνεδρίαση σήμερα για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε πώς θα διαρθρωθεί το κείμενο. Υπάρχει μία διαφορά σχετικά με αυτήν την εννέα θηρίδα, δηλαδή ε, να έχουμε και για τις λειτουργίες μια άλλη θηρίδα, να έχουμε δηλαδή δύο τύπων θηρίδες και για την ομάδα μου το βασικό πρόβλημα είναι στο παράρτημα όπου ορίζονται εννέα διάδρομοι. Εμείς ε, είμαστε εν αναμονή να έρθουν ε, άλλες πληροφορίες και βάσει αυτών των πληροφοριών που θα λάβουμε θα οριστικοποιήσουμε τη θέση μας. Αύριο στη συνεδρίαση που θα έχουμε ελπίζω ότι θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Αλκρόε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και από πλευρά σκιώδου του της ε, Δική μα ομάδα να πω κάποια πράγματα εγώ γιατί ο κύριος Λιμπεράτσκι απουσιάζει δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι πως ε, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη και το EMS ε, πρέπει να επεκταθεί αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης οι χώρες οι οποίες ε, θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα και να επενδύσουν πρέπει να υποστηριχθούν και κατά προτεραιότητα από την Κομισιόν. Κοιτάζοντας τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες του κυρίου Μαρινέσκου, αυτές οι οποίες έχει προτείνει ο συζητητής, ε, μπορούμε να τις υποστηρίξουμε και βεβαίω αναμένουμε μια πρόταση του Συμβουλίου σχετικά για να ξέρουμε να δούμε τι, ποια θα είναι η πραγματική κατεύθυνση στην οποία θα, θα κινηθούμε και θα έλεγα πως σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε οπωσδήποτε τον συγκητή και βεβαίως διμερώς θα, θα τα ξαναδούμε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κρέμερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Συνεργαστήκαμε έντονα, υποστηρίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες για τα τρία σημεία. Τώρα θα ήθελα να πω τα Για τις ε, διαταραχές ε, που υπάρχουν εκεί πέρα δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη θέση από το να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο πρόγραμμα που έχουμε. Βάσει δόγματος δεν μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητες σε άλλους και να καθυστερήσουμε κάποιους άλλους. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εάν μείνει στάσιμο ένα τρένο μετά από ένα ατύχημα και ο οδηγός, ο μηχανοδηγός πρέπει να κάνει διάλειμμα επειδή λύγει η βάρδιά του, είναι αδιάφορο το εάν είναι σε intercity, σε περιφερειακό τρένο ή σε φορτηγό τρένο πρέπει εντός των 15 λεπτών να φύγει το τρένο στο πρόγραμμα, αλλιώς θα κολλήσει όλο το σύστημα. Αλλιώς, ε, ακριβώς ειδικά για ατυχήματα, πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο η ευελιξία. Δεύτερον, για τη μία θηρίδα. Εάν δεν τα καταφέρουμε εδώ πέρα να το περάσουμε, τότε η όλη οδηγία δεν θα έχει κανένα νόημα θα, θα έχουμε χάσει μισό χρόνο, θα παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν, οπότε θέλουμε έναν συνομιλητή. Εν τω μεταξύ βεβαίως στις περιφέρειες οι υπηρεσίες της πόλης το έχουν κάνει αυτό ήδη. Και αν ε, δεν το καταφέρουμε εμείς εδώ πέρα δεν ξέρω ε, τι θα κάνουμε. Τέλος με τον διάδρομο. Δεν μπορέσαμε εμείς να εξηγήσουμε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε αυτός ο διάδρομος ή αυτή και οι έξι διάδρομοι του ERTMS. Γιατί μιλάμε για έξι, είναι δικαιολογία ή επειδή είναι περισσότεροι θα γίνουν γρηγορότεροι. Νομίζω πρέπει να περιοριστούμε νομίζω στους διαδρόμους. Οι διάδρομοι είναι διάδρομοι, δεν μπορείτε να γράφω συγκεκριμένη πορεία. και το ότι ο διάδρομος από τη Στοκχόλμη στην Κοπενχάγη πηγαίνει στο Αμβούργο, Ινσμπρουκ, ε, Νάπολη και Παλέρμο είναι λίγο αστείο δηλαδή. Εάν ήταν και η Φραγκφούρτη στη μέση το καταλάβαινα, αλλά γιατί πρέπει να πάει αυτός ο διάδρομος οπωσδήποτε μέσω Αμβούργου ενώ δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τούνελ ή γέφυρα ή οτιδήποτε και δεν θα χρηματοδοτηθεί ούτω ή άλλω για τα επόμενα 20 χρόνια και ξέρουμε τι γίνεται σε Αμβούργο, Ανόβερο και Βρέμι με τα μποτιλιαρίσματα, δεν έχει νόημα να κάνουμε την λύση που ακολουθούνται. Και βεβαίω ε, προ αυτή την κατεύθυνση, για μια αλλαγή δηλαδή σε αυτό το σημείο, θα είναι και οι τροπολογίε μα. Ευχαριστώ, Μάικλ. Grazie Presidente. Ευχαριστώ τον εισηγητή, έκανε εξαιρετική δουλειά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω μόνο δύο σημεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι λάθη. Στο παράρτημα 1, διάδρομος 5 δεν ανταποκρίνεται στη διαδρομή που έχουμε προχαράξει μεταξύ Βαλτικής και Αδριατικής και είναι η σύνθεση του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 23-25 και το 6 δεν ανταποκρίνεται επίσης με το χάρτη του PP6. Τώρα άλλη παρατήρηση για τις προτεραιότητες. Εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να ξανα ορίσουμε ορισμένες τροπολογίες για τις ώρες εχμής, ε, τις οποίες ε, είχε υποβάλει ο κύριος Μπερτίνη και τις πέρασε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και τις έκοψε μετά το Συμβούλιο. Αυτό το λέμε για να δώσουμε προτεραιότητα στους επιβάτες ε, και όχι στα εμπορεύματα. Όταν μιλάμε εμείς για κίνηση, οι κανόνες προτεραιότητας δεν πρέπει να εφαρμόζονται κατά τις ώρες εχμής όπως αυτές έχουν οριστεί στο, κάθε κράτος μέλος. Παρακαλώ επίσης τον εισηγητή να εξετάσει το θέμα της διαλουργικότητας και της ε, ε λειτουργίας ε, της σιδηροτροχιάς ε, για τα διάφορα τρένα επιβατικά, εμπορικά κλπ υψηλή ταχύτητας. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνεται είναι αρκετά δύσκολος προς τη διαχείρισή του. Κύριο Μπαχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Θα ήθελα συνολικά να στο όσο ευπρόσδεκτη την πρωτοβουλία, ιδιαίτερα για τους ε, ε, διαδρόμους για τη μεταφορά φορτίων που θα βελτιώσει σημαντικά και τους, τις μεταφορές αλλά και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, γιατί όσε δηλώσει και να κάνουμε και στι πολιτικέ πρωτοβουλίε και να λαμβάνουμε για να μεταφέρουμε το φορτίο στο σιδηροδρόμο, χωρί αυτέ τι σημαντικέ ε, βελτιώσει ω προ την ποιότητα, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το σημείο εκκίνηση επίση είναι για μένα μια καλή ιδέα μια καλή πρωτοβουλία. Ε, ασφαλώς χρειάζεται η πολιτική ανεξαρτησία, που πρέπει να εξασφαλίσουμε, και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή κοινή προσπάθεια, ώστε οι εταιρείες μεταφοράς φορτίου να ε, τηρήσουν τις πιο αυστηρές και σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, να υιοθετήσουν τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας στο ε, σιδηροδρομικό του υλικό, στο τροχαίο υλικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Η αρχή της, της δημιουργίας ενός διαδρόμου ε, είναι να μπορέσει να επιταχύνει την μεταφορά των εμπορευμάτων ε, και, με, και βοηθώντας τις συνδυασμένες μεταφορές και τους επιβάτες βέβαια. Αλλά ο βασικός λόγος δημιουργίας αυτών των διαδρόμων είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών του τομέα της ε, μεταφοράς εμπορευμάτων. Το να δώσουμε εμείς προτεραιότητα στη διαμετακόμιση των επιβατών ε, αντιβαίνουμε στο πνεύμα της ε, δημιουργίας της ίδιας της ε, οδηγίας. Εμείς θα πρέπει να ξαναβάλουμε αυτό το σημείο στην έκθεση και, μετά, και αυτό που είπε και ο κύριος Μπάχ, ότι θα έχουμε ίσους όρους ασφάλειας στις ε, μεταφορές ε, εμπορευμάτων και επιβατών. Αλλά για τα τρένα όμως τα ίδια, δηλαδή για την υποδομή, ε, είναι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και όσο πιο πολύ εμείς ε, συγχαίουμε τη μεταφορά εμπορευμάτων με την ε, ε, μεταφορά επιβατών, τότε θα υπάρχει πάντοτε πρόβλημα και με τα θέματα ασφάλειας, αλλά και με τα θέματα του, των υποδομών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση. Δεν ήταν εύκολη. Βέβαια, ευχαριστώ και τον προηγούμενο συγκεκριτή για την προηγούμενη εργασία του. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Ε, μιλούμε για διαλειτουργικότητα, θέλουν περισσότερες μεταφορές ε, στη σιδηροτροχιά. Πλην όμως δυστυχώς στην Ευρώπη δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ρυθμίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να ε, εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη εξού και δεν προώθησαν ε, τις ρυθμίσεις για τις μεταφορές φορτίων με βάση το, την αντίστοιχη νομοθεσία για τα πρόσωπα, για τους επιβάτες δηλαδή τα κράτη-μέρη. Είναι κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε στη Γερμανία πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους περιβαλλοντικούς. Να διευκολύνουμε τη χρήση του σιδηροδρόμου και από τους επιβάτες αλλά και για τα φορτία. Αυτό λοιπόν θέλουμε να προωθήσουμε. Θέλουμε δηλαδή τις ε, καλύτερες δυνατές λύσεις ε, για τα φορτία και βέβαια λύσεις οι οποίες να είναι εφαρμόσιμες στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια λεπτή ισορροπία την οποία ασφαλώς έχει εξασφαλίσει η συνεργασία με τους κοινούς και θα εξασφαλίσει ο εισηγητής μας. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Σέπινγκ. Εντάξει, καλώς. Ε, για την Κομισιόν μετά, ο κύριος Καστελέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω γενικά αυτή τη στιγμή. Στην αρχή της δεύτερης ανάγνωσης αυτής της νομοθετικής πρότασης θα θέλαμε να επαναλάβουμε ακόμη μία φορά με έντονους όρους την ε, οικονομική και πολιτική σημασία της πρότασης αυτής γνωρίζετε πως η οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα τις εμπορευματικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων καθώς ο παραδοσιακός πελάτης είναι η βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, χημικά, μέταλλα, χάλιβας και όλα αυτά έχουν μειωθεί κατά πολύ από το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στο τέλος του 2009 έχουμε μία επιστροφή στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 90. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε πως υπάρχουν κάποια βασικά διδάγματα που πρέπει να αντληθούν για να αναζωογονηθεί ο τομέας, καθώς πρόκειται για έναν τομέα διεθνή και πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ε, απαραίτητος παράγοντας βέω είναι η ποιοτική υποδομή ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό το ζητούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Οι καλές διεθνείς υποδομές είναι βασικός όρος για την ανταγωνιστικότητα πολλών τμήματων ε, των σιδηροδρομικών μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών. Οπότε είναι ε, Βεβαίω, για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν επίση όρει τα άλλα μέσα μεταφορά. Πριν μπω σε άλλε λεπτομέρειε, θα ήθελα να απορρίψω πριν περάσουμε και στην έκθεση του Συμβουλίου κάποιες αμφιβολίες που ακούστηκαν και βλέπουμε πως οι ίδιε αμφιβολίες επανεφανίζονται και εδώ πέρα. Κάποιοι είναι κατά αυτής της πρότασης γιατί πιστεύουν πως ε, θα βλάψει την ε, μεταφορά επιβατών και ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα απορρίπτει αυτά η Κομισιόν και θεωρεί πως είναι λανθασμένη η ερμηνεία της πρότασης. Η εμπειρία δείχνει πως η δυναμικότητα των σιδηροδρόμων μπορεί να καταφέρει να εξυπηρετήσει και επιβάτες και φορτίο. Δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται οι μεταφορές εμπορευμάτων τους επιβάτες, αλλά τις οδικές μεταφορές. Κάποιοι άλλοι είναι υπέρ του status quo λέγοντας πως ε, πρέπει να επικρατήσουν οι δυνάμεις στις αγορές, αλλά βεβαίως αυτοί έχουν προνομιούχες σχέσεις με όσους διαχειρίζονται τις εθνικές υποδομές και εμείς θέλουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, διάφανο και προβλέψιμο δίκτυο, το οποίο θα είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να επενδύσουν. Η νομοθετική πρόταση που εξετάζουμε σήμερα περιέχει τα στοιχεία ανάπτυξης ποιοτικής υποδομής ε, των σιδηροδρόμων και αυτό συμπεριλαμβάνει και την συνεργασία των διαχειριστών σε επιχειρησιακά ζητήματα και ζητήματα επενδύσεων, την αξιοπιστία επίσης ε, των υποδομών, τη σχέση μεταξύ του δικτύου και των υποδομών αποθήκευσης και τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των διαφορετικών εταιριών. Επίσης, το Συμβούλιο βασίζεται στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως κάποια στοιχεία έχουν κάπως αποδυναμωθεί, όπως παραδείγματο χάρη διαδικασία επιλογής διαδρόμων, η συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών της υποδομή Επιπλέον, κάποια άλλα στοιχεία όπως ε, το να υπάρξει κάποιος ετών ο οποίος δεν θα έχει προεγκριθεί ή το να απευθυνόμαστε σε μία μόνη υπηρεσία έχουν αφαιρεθεί εντελώς. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν εξακολουθεί να θεωρεί πως η κοινή θέση του Συμβουλίου μπορεί να είναι σύμφωνη με το σκοπό της αρχικής πρότασης της Κομισιόν αναμένουμε τώρα μια γρήγορη υιοθέτηση αυτής τη νομοθετικής πρωτοβουλίας και κατά τη διάρκεια της δεύτερη ανάγνωσης ο γενικός στόχος της Κομισιόν λαμβάνεται υπόψη και υπογραμμίζουμε το επίπεδο φιλοδοξίας ε, του νομοθέτη που είναι σύμφωνο με αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Marinescu. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Ε, thank you, ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως έλεγα νωρίτερα, η πρόταση του Συμβουλίου προσφέρει ένα νέο στοιχείο. Το παράρτημα με το οποίο αμέσως λαμβάνεται η απόφαση για ορισμένους ε, διαδρόμους και συμφωνήσαμε να την υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερος τους ε, σκιώδης ηγητές και όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν ε, στις προτάσεις μου μέχρι τώρα. Συμφωνήσαμε διότι θεωρούμε ότι προχωρούμε έτσι σε μια ταχύτατη υλοποίηση της έκθεσης. Εάν λοιπόν συμφωνήσουμε ως προς τις κύριες γραμμές των διαδρόμων και εφόσον ε, πληρούν και οι διάδρομοι τα κριτήρια, μπορούν να ε, μετατραπούν σε διαδρόμους για φορτίο, όπως άλλωστε θα κρίνουμε με την συνάντηση που σκοπεύουμε να οργανώσουμε σύντομα και λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των συναδέλφων όπως του κ. Κατησιάνη και όλων των άλλων που μίλησαν εδώ με όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν τους ε, διαδρόμους και που θα περιλάβουμε στην πρότασή μας. Στα γραφειοκρατικά τώρα. Εδώ ε, πρόκειται για διάδρομο φορτίου και όχι για τροχαίο υλικό, ούτε για διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι κάτι το αυτονόητο όταν προσπαθούμε να χαράξουμε ε, μια τέτοια εμβέλεια καινοτομία. Δηλαδή πρέπει να εισάγουμε και νέα στοιχεία σε επίπεδο θεσμικό. Θα χρειαστεί και αυτό λοιπόν όντω. Θα χρειαστούν δύο συμβούλια συντονισμού. Το ένα με τα κράτη-μέλη και το άλλο με τους ε, παρόχους υποδομών, με τους χειριστές δηλαδή υποδομών σε επίπεδο εθνικό. Αλλά πιστεύω ότι και τα δύο θα διευκολύνουν ιδιαίτερα και θα βελτιώσουν ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των διαδρόμων. Και επίσης πιστεύω ότι όταν μιλούμε για προτεραιότητα δεν μπορούμε σε συνήθεις όρους να δίνουμε προτεραιότητα στο φορτίο έναντι του, ε, της μεταφοράς επιβατών ή αντίστροφα να πούμε ότι οι επιβάτες πάντα πρέπει να έχουν την προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να μιλούμε με τέτοιου όρου. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύσει ώστε να επιτρέψουμε την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ε, η ροή και των δύο τύπων μεταφορών. Εάν όμω προκύψει πρόβλημα στι μεταφορέ, διαταραχή δηλαδή στι μεταφορέ, τότε θα πρέπει να έχουμε κάποια λύση έτοιμη. και νομίζω ότι ε, η λύση η οποία θα διευκολύνει την αποκατάσταση της ομαλής ροής ε, των μεταφορών θα είναι και η καταλληλότερα. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει αρκετές προτάσεις, αλλά τώρα θα πρέπει να δούμε πολύ πιο συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι απαντήσει θα δίνει όταν κάποιο καταθέτει αίτηση για δημιουργία ενό διαδρόμου, που θα πρέπει να απαντά μέσα σε ένα εξάμεινο η Επιτροπή και η υλοποίηση να προχωρήσει μέσα σε δύο ή τρία χρόνια. Έτσι λοιπόν τότε θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι για την υποστήριξή σας και πιστεύω ότι έχετε δυνατό... να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τροπολογίες μέχρι τις 22-23 Μαρτίου, τις οποίες θα τις εξετάσουμε 3 Μαΐου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 4 Μαΐου και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο, για να σας δώσω το πρόγραμμα. Ωραία. Διακόπτεται τώρα η συνεδρίαση μέχρι τις 3 παρα 10 όταν θα γίνει η ψηφοφορία για την ασφάλεια της αεροπορίας. Οπότε μπορείτε όσοι δεν έχετε τις κάρτες σας να πάτε να τις πάρετε. 15 και 50 λοιπόν για την ε, ψηφοφορία. Δεν μπορώ να το φέρω πιο μπροστά, είναι ψηφοφορία για σας. Hey, ladies and gentlemen, can we take our seats? The... Κυρίες και κύριοι, καθίστε. Λοιπόν, είναι 4 παρα 10. Λοιπόν, σχέδιο έκθεσης για τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, η έκθεση Lightfried. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ματίας, να σας ενημερώσω πως η τροπολογία υπαριθμών 69 αποσύρεται. 69 του κυρίου Μαρινέσκου. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Ξεκινάμε άρθρο 1, παράγραφος 1, τροπολογία 43 Μαρινέσκου και αυτή έχει αποσυρθεί. Οπότε 46, 47, 49 που είναι ταυτόσιμες των κυρίων Κοχ, Κουν, της κυρίας Αγιάλα Σέντερ και Άλβαρες. Υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτονται. Ερτούγ 50 ήταν ταυτόσημιο, 45 Ήταλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 Ντεβεϊράκ αποσύρεται. 7 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 48 άρα καταπίπτει. Μετά 51 η κυρία Γιάλα Σέντερ και ο κύριος Άλβαρες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 53 στο άρθρο 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 αποσύρεται 54 χωριστή ψηφοφορία του κυρίου Μανέσκου το πρώτο μέρος είναι όλοι οι 54 χωρί τις λέξεις serving the same city conurbation το δεύτερο τμήμα συμπεριλαμβάνει αυτή τη διατύπωση Πρώτο τιμά χωρίς αυτές λέξεις υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτό. Οπότε, το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 2, Β, Α, νέο 8 του εισηγητή και 55 του κυρίου Φέρμπερ είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η παριθμόν 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 Δανέλης προσθήκη υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 2, δέλτα άλφα νέο 10 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3α νέο 11 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Οπότε 57 καταπίπτει. 12 του εισηγητή υπέρ κατά άποχες δεκτή 13 υπέρ κατά άποχες δεκτή 14 υπέρ κατά άποχες δεκτή συμβιβαστική τροπολογία α στο άρθρο 5 παράγραφος 2α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κύριε Λάιχτφριντ, εγώ αποσύρω την δική μου την 15. Ε, Επιτρέπετε, μπορείτε να την αποσύρετε, οπότε 58, 59, 60 και 61 είναι ταυτόσιμες υπέρ ο εισηγητής δεν είμαι σίγουρος κύριε πρόεδρε αλλά εάν α ναι όχι όχι με συγχωρείτε εντάξει ναι ναι έχει αποσυρθεί άρα δεν καταπίπτουν 58, 59, 60, 61 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτές 16 εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 62 άρθρο 4 παράγραφος 4 η κυρία Γιαλασέντερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 Αλμπερτίνη υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Νομίζω πως έχει καταπέσει αλλά θα ήθελα να το δω. 63 του κυρίου Αλμπερτίνη. Άρθρο 4, 4α. Άρχιδη σοφορία. Πέρας. 19 υπέρ, 19 κατά. Οπότε απορρίψετε. Ναι, δεν, δεν ξαναγίνεται Ματίας, συγγνώμη. Έπρεπε να γίνει σωστά από την αρχή όταν είναι τόσο τσιματσίμα. Όχι, όχι, δεν, δεν πρόκειται να επαναλάβω την ψηφοφορία επειδή είναι ακριβώς, επειδή είναι ισοψηφία. Ε, ναι, αλλά δεν δουλεύει το μηχάνημά της. Δεν, δεν γίνεται τώρα εκ των υστέρων. Προτείνω να την ε, επανυποβάλλετε στην Ολομέλεια. Να την επα... Ναι, αλλά πώς ψήφους έχουμε στο ΕΛΚ αυτή τη στιγμή, λέει ο κύριος Γκρός, σε αυτή την ψηφοφορία. Ε, δεν ξέρουμε τώρα γιατί το σβήσαμε. Όχι, μπορείτε βεβαίως να το έχετε. Η πρότασή μου, λέει ο πρόεδρο, εάν επιμένετε τόσο για αυτήν την τροπολογία, να την ξαναφέρετε στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια θα αποφασίσει. Εάν το κάνω αυτό κάθε φορά που είναι ισοψηφία, θα, κάποιος θα λέει δεν δουλεύει το μηχάνημα. Ναι, αλλά αν κάποιο έχει πρόβλημα, το ξέρει αφού ψηφίσει, αφού προσπαθήσει να ψηφίσει. Θα σας πω λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μία δοκιμή Μία δοκιμή τη ψηφοφορία. Δεν θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Μπορούν να ψηφίσουν όλοι. Απλά δοκιμάζουμε. Δουλεύει το μηχάνημά σας, κυρία συνάδελφε. Ναι, ναι δουλεύει. Οπότε το αποτέλεσμα ισχύει. Άρθρο 4, υπαριθμό 19. Ναι, με συγχωρείτε, όχι. Για κάτι άλλο. Εγώ έχω την κάρτα μου εδώ πέρα. Στην κάρτα μου λέει το δικό μου όνομα και ο υπολογιστή λέει Smith. Εάν έχετε κάποιον Smith λοιπόν είμαι εγώ. Ναι ξέρουμε πως Smith είναι Στέρξ στα φλαμανδικά. Ματίας. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να ελέγξετε πόσοι ψηφίζουν σοσιαλιστές αυτή τη στιγμή. Σοσιαλιστές. από ό,τι βλέπουμε είναι εντός της ποσόστοσής τους. Όχι είναι ένας παραπάνω. Αυτό έδειξε το μηχάνημα. Όχι. Αντιθέτως πράσινη είναι ένας παραπάνω. Δεν θέλω να επαναλάβω την ψηφοφορία, σας είπα γιατί, γιατί έτσι δημιουργείται προηγούμενο για ολόκληρη τη θητεία. Κάθε φορά που είναι τσίμα τσίμα η ψηφοφορία θα λέει κάποιος το μηχάνημά μου δεν δουλεύει. Αν δεν σας αρέσει η απόφαση του Προέδρου θα πρέπει να την προσβάλλετε αλλού. Προχωράμε, μπορείτε να επανυποβάλλετε την τροπολογία στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια θα αποφασίσει. Άρθρο 4, παράγραφος 4, β, 19. Επ' αυτού του ζητήματος. Ναι, επειδή ο κύριος Γκρός μετράει 12 σοσιαλιστές, αλλά μόνο 11 ψηφίζουν, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, κοιτάξτε, το μηχάνημα δεν μας δείχνει ότι είναι παραπάνω οι σοσιαλιστές. Μόνο οι πράσινοι. Και αυτό το λάβαμε υπόψη. Τροπολογία 19 σε 3 μέρη χωριστή ψηφοφορία ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Πρώτο τμήμα, μία εποπτεύουσα αρχή κράτους μέλους, δεύτερο μέρος ε, διεξάγεται από αυτή την αρχή, ε, τρίτο μέρος οι διαδικασίες μέχρι και διάφανο. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές δεκτό 20 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ένας πράσινος παραπάνω, κύριε Κράμερ. Είναι όλοι εντάξει με τα μηχανήματά τους, με τα δακτυλάκια τους, όλοι εντάξει. Πέρας της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται, 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρθρο 5, παράγραφος 1, β, α, νέο, 21, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 22 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 υπέρ. κατά αποχές δεκτή. 66 Μαρινέσκου σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 καταπίπτει. Οπότε είμαστε στο 5-2 εισαγωγή, 25 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 67. Ο κύριος Γκρόσο επί της Ναι κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εάν συμφωνείτε να σας ζητήσω να ξαναδεί, να μας εξηγήσει εδώ πέρα η συντάκτη στην τροπολογία. Δεν καταλαβαίνουμε εδώ πέρα τι εννοούν στο ΕΛΚ. Σύντομα, εάν μου επιτρέπετε, η 67 της κυρίας Ένης Πλασέρτ. Κυρία Χένις Πλάσσερτ, υπάρχει κάποια σύγχυση. Τι θέλετε να μας πείτε εδώ πέρα. Ξέρω πως η συγητής έχει προτείνει να καταψηφίσουμε μετά την γνωμοδότηση της Κομισιόν, αλλά επιμένω σε ένα συν. Δεν έχω τώρα το επεξηγηματικό σημείωμα αλλά αφορά την αποτελεσματικότητα που συνδέεται με την ασφάλεια. Οπότε ζητώ το, από το ΕΛΚ να ψηφίσει εδώ μαζί με τους φιλελεύθερους. Μάλιστα. Δεν ξέρω εάν σας ικανοποιεί αυτή η εξήγηση, αλλά είναι μία εξήγηση εν πάση ε, Μπράιαν, δεν θα κρίνεις εσύ. Δεν θα κρίνω εγώ, πράγματι λέει ο πρόεδρος. σύντομα. Κοιτάξτε, να πιούμε, να πιούμε ένα φλιτζανάκι καφέ, να μου εξηγήσετε, αλλά μέχρι να μου το εξηγήσετε είμαι κατά. Μάλιστα, 67 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 καταπίπτει, 69 έχει αποσυρθεί. 70 καταπίπτει λόγω της 29, οπότε φτάνουμε στην 30, άρθρο 6, παράγραφος 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 71 Hennis Πλάσσερτ υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αυτή νομίζω ήταν πιο Σε 73 χένι Πλασέρτ υπέρ. Ε, τι σου Μπράιαν. 73 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Την 73 της κυρίας Χένις Πλασέρτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 26 υπέρ 14 κατά δεκτή, άρα η 74, 74 74 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε 74 του κυρίου Μαρινέσκου. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. τα πίπτη. 20 υπέρ, 20 κατά. 75 Ζασάντα υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε και αυτό, παρακαλώ, 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 20 κατά και αυτή απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 ζασάντα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Άρθρο 8, 1α31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 τρεμόσα ή μπαλσέλς υπέρ κατά Εποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 τρεμόσα υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτεί. 36 Αλμπερτίνη υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας ένα τώρα ε, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 37 Λίχτενμπέργκερ, Κλάμερ και Τιράντ υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να υπαλληθεύσουμε, Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά πρέπει να ελέγξουμε 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 16 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται 38 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές με την ίδια διαφορά απορρίπτεται 2 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 πίπτη 40 έχει αποσυρθεί 41 προσθήκη υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας 5-3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 42 για Λασέντερ Άλβαρες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. τελική ψηφοφορία. Η νομοθετική πρόταση, όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 36 υπέρ, κανείς κατά 4 αποχές γίνεται δεκτή και το νομοθετικό ψήφισμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 34 υπέρ, 5 αποχές, κανείς κατά δεκτό. Συγχαρητήρια κύριε Λάιχτρη. Next item on the agenda. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μάικλ Θέλω απλώ να πω, Πρόεδρε, μια και είπατε νωρίτερα ότι ψήφισε ένα περισσότερο από του πράσινου. Εγώ βρήκα μόνο λοιπόν τρει πράσινου. Τρει ψήφου έχουμε και δεν καταλαβαίνω πού βρήκατε την τέταρτη ψήφο. Και δεν έχω και δύο κάρτες για να ψηφίζω. I can only tell you, Mr. Kramer, what a... Κύριε Κράμερ, εγώ το μόνο μπορώ να πω είναι αυτό που βλέπω στην οθόνη της τηλεόρασης, που μου δείχνει μία ψήφο παραπανίσια. Άλλο τίποτα δεν ξέρω να πω. Μα δεν αμφισβητώ την, ε, το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία, λέει ο κύριο Κράμερ. Απλώ μην μου λέτε ότι ψηφίσαμε 4 αντί για 3. Μήπως ο κύριος Σμιθ ε, ε, εκ Φλάνδρας. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα ελέγξουμε. Ειδικά όταν είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά στενά, πρέπει να ελέγχουμε. Θα κάνουμε την επαλήθευση λοιπόν. Το επόμενο θέμα που έχουμε είναι η έκθεση για την ασφάλεια των ενέργειων μεταφορών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την προστασία των θυμάτων ατυχημάτων και θα ήθελα να καλωσορίσω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση εκπροσώπους της ΦΕΝΒΑΚ, της Ομοσπονδίας δηλαδή θυμάτων αεροπορικών ατυχημάτων. Πρόκειται για οικείους θυμάτων αεροπορικών δυστυχημάτων της ε, ε, πτήσης 447 από το Ρίο Ντετζανέιρο στο Charles de Gaulle της Spanair και άλλων ε, γνωστών σε όλους μας ε, αεροπορικών δυστυχημάτων. Λυπούμαστε βαθύτατα για ε, τα, την απώλεια των αγαπημένων σας προσώπων και είσαστε βέβαια ευπρόσδεκτοι εδώ στην συνεδρίασή μας. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Ντεβεγάκ να κάνει την παρουσίαση της εκθεσής της. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την προετοιμασία του εγγράφου εργασία, το οποίο έχουμε διανύμει, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλούς εκπροσώπους ε, από τον τομέα της, ε, των ενέργειων μεταφορών, από την ΕΖΑ, την Airbus, ε, τις, εταιρεία αεροπορικών μεταφορών και τις Ομοσπονδίες Οικείων Θυμάτων των Αεροπορικών Δυστυχημάτων, τους οποίους και καλωσορίζω εδώ και ευχαριστώ ιδιαίτερω για την παρουσία τους. Επίσης είχα μαζί με εσάς, Πρόεδρε, ε, όπως και με συναδέλφους της ΤΡΑΝ, την ευκαιρία να, να επισκεφθώ το, τη Βρετανική Υπηρεσία για την ε, διαλεύκανση αεροπορικών δυστυχημάτων και το αντίστοιχο γαλλικό αργότερα. Βλέπω λοιπόν από όλα αυτά ότι μπορεί να είναι πολύ πλήρης και να έχει αρκετά τεχνικό χαρακτήρα η έκθεση επιτροπή, αλλά πάντω έχει τεράστια σημασία για τι εναερίε μεταφορέ και την ασφαλειά του. Έχω λοιπόν επιλέξει διαφορετικέ λύσει μέσα στο έγγραφο εργασία μου και θα ήθελα πολύ να σα αναφέρω. Καταρχά, όσον αφορά το δίκτυο των αρχών διερεύνηση. Οι εθνικέ υπηρεσίε κίνδε στο επίκεντρο τέτοιου είδου ε, ερευνών και οι αρμόδιες αρχές με τη δουλειά τους είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να προσδιορίσουν τις αιτίε ενός δυστυχήματος και να αποτρέψουν στο μέλλον την επαναλήψή του. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να τους προσφέρουμε το κατάλληλο πλαίσιο, έτσι ώστε την έρευνά τους να την αναπτύσσουν με τρόπο απόλυτα ανεξάρτητο και να εντοπίζουν τα κενά, τα προβλήματα ως προς την ασφάλεια. Προτείνουμε λοιπόν τη θέσπιση ευρωπαϊκών γραφείων, ε, έτσι ώστε να συντονίζονται καλύτερα οι εργασίε των εθνικών γραφείων. Όμω η Επιτροπή δεν έχει αναπτύξει την ιδέα αυτή επαρκώ. Και εγώ θα ήθελα να προχωρήσω λίγο περισσότερο και να προτείνω συγκεκριμένα προσδιορισμό τη αποστολή αυτού του δικτύου, του ευρωπαϊκού δικτύου, που θα προσφέρει με, την, με τον τρόπο αυτό την προσθέμενη του αξία προ την ασφάλεια των αέριων μεταφορών. Αντίστοιχα, έχουμε στελεστέ μεταφορέ μια υπηρεσία, ένα δίκτυο μάλλον διερεύνηση των ε, ναυτικών ε, ατυχημάτων, ναυαγίων κτλ. Ε, και άρα αντίστοιχα για τις ενέργειες ε, μεταφορές θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις βέλτιστες ε, πρακτικές, για μια συνδυασμένη δραστηριότητα στην έρευνα, ε, και τους ελέγχους. Πρέπει όμως να σημειώσω ότι το δίκτυο δεν θα αποτελέσει νέα υπηρεσία, δεν θα έχει νομική προσωπικότητα, ούτε θα αποτελέσει ένα νέο και πρόσθετο όργανο. Απλώς βελτιστοποιεί τις υφιστάμενες δυνατότητες και την εργασία και την αποτελεσματικότητα του κάθε χωριστού γραφείου ή υπηρεσίας Επίσης, εδώ υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια αυτό το δίκτυο. Απλώ θέλουμε να το πλαισιώσουμε καλύτερα και να οργανώσουμε την αποστολή του κατά τρόπο ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διερεύνηση. Δεν υποκαθιστά, ούτε στόχο έχει να υποκαταστήσει τις ε, υπηρεσίες. Ε, απλώς προσπαθεί να βελτιώσει τις επιδόσεις των πάντων και τα 27 κρατη με τι 27 του υπηρεσίε, να μπορέσουν να συντονιστούν καλύτερα για πιο αποτελεσματική διερεύνηση. Θα αποτελέσει δηλαδή το μέσο για την παραπληρωματικότητα των λειτουργιών και εργασιών των υπηρεσιών των κρατών μελών. Έτσι ώστε να έχουμε 27 αποτελεσματικέ υπηρεσίε διερεύνηση στα κράτη-μέλη. Άρα έχει τεράστια πολιτική σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η πρόταση και καθώ μάλιστα το Συμβούλιο προσπαθεί να το ε, απογυμνώσει από τις αρμοδιότητες του και πάνω απ' όλα από την ουσία του, πράγμα το οποίο θα σήμαινε ότι θα ειστρέφουν τα πάντα σε μια ε, μπεμονωμένη δράση των υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προσδορίσουμε και το πεδίο δράση και την ουσία αυτού του δικτύου μέσα από τον κανονισμό. Και εδώ πρέπει να επιμένουμε ιδιαίτερα αυτό το Συμβούλιο όταν είστε αντίθετα με τι δικέ μα προτάσει. Επίση, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Αεροπορία, ο οποίο αντικαθιστά εδώ και αρκετά χρόνια τα κράτη-μέλη ω προ την αρμοδιότητα πιστοποίηση των αεροσκαφών στην κοινότητα και άρα πρόκειται για μείζωνα παράγοντα τη ασφαλή εναέρεια κυκλοφορία. Άρα λογικό είναι αυτό ο οργανισμό να παρεμβαίνει στι έρευνε, ε, στη διερεύνηση των ατυχημάτων και να βοηθάει τους ερευνητέ. Πλην όμω ε, και ενώ τα γραφεία διερεύνηση, οι υπηρεσίε διερεύνηση των κρατών μελών έχουν μακρά εμπειρία και συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, που μερικέ φορέ δεν πάγεται και στο Διοπουργείο, δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Αεροπορία, που είναι πρόσφατο θεσμό πρόσφατη υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν έχει, δεν έχει αναπτυχθεί η συνήθεια συνεργασίας ε, με τις εθνικές υπηρεσίες διερεύνησης και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε και συγκρούσεις προς το ποιο είναι ο αρμόδιος για ποια έρευνα, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα προς εξέγον της έρευνας. Εμεί λοιπόν θέλουμε εδώ να θεσπίσουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, χωρί όμω αυτέ οι δραστηριότητε να σημαίνουν για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό τη δυνατότητα να επηρεάσει την έρευνα για την ασφάλεια ή να ε, αναπτύξει παράλληλη έρευνα. Δηλαδή, ναι, μεν έχει την πιστοποίηση Αυτό ο οργανισμό, ταυτόχρονα όμω δεν μπορεί και να κρίνει τα αποτελέσματα αυτή τη πιστοποίηση, Δεν μπορεί δηλαδή να είναι και κριτή και ε, διάδικος. Και γι' αυτό και για να προσδιορίσουμε καλύτερα το ρόλο του οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στην έρευνα, θέλουμε σαφέστερη διατύπωση του άρθρου 13 του αντίστοιχου νομοθετήματος. Θα προτιμούσα λοιπόν, για να μην υπάρχουν παρεμηνίε ω προ την περιγραφή του ερευνητή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουν μια σαφή διατύπωση, έτσι ώστε να μην μπορούν να αμφισβητηθούν οι δραστηριότητε του από κανέναν και γι' αυτό θα πρότεινα τη λέξη σύμβουλο ε, για την αρχή πιστοποίηση. Έτσι λοιπόν ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίηση θα χαρακτηρίζεται ω σύμβουλο και αυτή θα είναι και η συμμετοχή του στι ε, δραστηριότητε διερεύνηση των ατυχημάτων και θα δίνει τι συμβουλέ του όπω ορίζεται στο παράρτημα υπερθυμών 13. Ξέρω ότι η η συμμετοχή του, οργανισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για σας έχει μεγάλη σημασία, αλλά για μένα το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό τόσο όσο νομικό, δηλαδή πρέπει να βρούμε την κατάλληλη περιγραφή και το κατάλληλο πλαίσιο, χωρίς να υπερβάλλουμε τη σημασία του ζητήματος αυτού, γιατί υπάρχουν πολλοί άλλα πολύ πιο σημαντικά μέσα στο κείμενο. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να δείξω είναι ο συντονισμός των διερευνήσεων και της ε, νομικής διαδικασίας, δικαστικής διαδικασίας. Ε, όντως μπορεί να υπάρχουν μία ή και περισσότερες δικαστικές διαδικασίες παράλληλα με τη διερεύνηση. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα παραμείνει ανεξάρτητη η διερεύνηση ασφάλειας. Ότι οι ελεγκτές θα μπορούν να εξετάσουν οτιδήποτε πιστήρια υπάρχουν χωρίς να χρειάζεται να λάβουν από κάποιον δικαστή τη σχετική άδεια. Πράγμα το οποίο όμως δεν είναι εξασφαλισμένο πάντοτε. Μια σημαντική επίσης ε, διάσταση είναι η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, δηλαδή τα στοιχεία που συλλέγουν οι ε, ελεγκτές κατά τη διακρύβωση των συνθήκων. Αυτά έχουν να κάνουν δηλαδή είτε με το μαύρο κουτί, είτε με την επαφή και τις συνεντεύξεις με τους ε, εναέρους ελεγκτές, είτε με άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος. Εάν ε, ε, κάποιος φοβάται να δώσει απαντήσεις στους ε, ερευνητές για, λόγω του φόβου ότι μπορεί κάποια στιγμή οι δηλώσεις του να εμπλακούν μέσα σε ένα δικαστικό φάκελο και να βρεθεί υπόλογος ενώπιον της δικαιοσύνης, προφανώς δεν μπορεί να γίνει σωστά η διερεύνηση των λόγων του ατυχήματος. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε και να παρεμποδίσουμε τη λειτουργία της δικαιοσύνης και να μην επιτρέψουμε και στις οικογένειες των θυμάτων να δουν άπλετο φως να ρίχνεται στο ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθεί κατάλληλη ισορροπία, η χρυσή τομή μεταξύ των δύο αυτών βασικών επιταγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει την προστασία ορισμένων προσωπικών στοιχείων ή πληροφοριών με τη δυνατότητα όμως εάν υπέρτατη ε, έννοια δημόσιου συμφέροντο απαιτεί να αποκαλυφθούν τα στοιχεία αυτά. Όμω αυτή η υπέρτατη έννοια του δημοσίου συμφέροντο διαφέρει από το ένα κράτο μέλο στο άλλο και πολύ συχνά όταν το ατύχημα ε, οδηγεί σε θάνατο, όπως δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει, ε, αναγνωρίζεται ότι επικρατεί η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και άρα δεν προστατεύονται παρκώς οι ευαίσθητες πληροφορίες στα προσωπικά δεδομένα. Εγώ προτείνω λοιπόν μια καλύτερη προστασία από αυτήν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνω ό,τι έχει να κάνει με την διαπίστωση των στοιχείων και την ανάλυση των πιστηριών να διαβιβάζεται στη δικαιοσύνη, αλλά οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με προσωπικά στοιχεία όπως οι συνεντεύξεις με τους παθόντες ή με τους εμπλεκομένους να παραμένουν απόρριτα. Και εδώ το, γράφω, έχουμε αυτό καταγράψει στο σημείο 15 παράγραφος 2 με ε, απόρριτα τα στοιχεία που καταγράφονται στο 15.2. Η η υπηρεσία η οποία έχει την ε, επεξεργασία των στοιχείων όπως και η Επιτροπή θεωρώ ότι δεν είναι παρκής η ε, προστασία των δεδομένων και η δική μου η πρόταση είναι πιο σύμφωνη με την γνωμοδότηση αυτής της υπηρεσίας, του οργανισμού καλύτερα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μένα, το πιο σημαντικό για, κατά την απόψή μου, είναι τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικείων τους. Έχουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα λοιπόν με τον κατάλογο των επιβατών με την κατάσταση επιβατών. Εδώ πρέπει να ορίσουμε, πιστεύω, σε ε, προθεσμίε, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να περιπέσουμε σε καταχρήσει, όπω ήταν σε πρόσφατα ε, ατυχήματα με προβλήματα σημαντικά για τους συμπολίτε μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η εταιρεία να έχει την υποχρέωση να ε, παρουσιάσει την κατάσταση επιβατών μέσα σε μία ώρα από, την, ε, από το ατύχημα. Θα συμφωνούσα εγώ καταρχήν βεβαίω, αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι πρέπει να είναι και ρεαλιστικές οι προθεσμίες. Μην ξεχνάμε ότι οι υπηρεσίε δεν έχουν πάντοτε στο αεροδρόμιο από το οποίο έχει απογειωθεί το αεροπλάνο μόνιμο προσωπικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αεροδρόμια τα οποία κλείνουν τη νύχτα. Και άρα πάνω απ' όλα, απαραίτητο για μένα είναι να υπάρχει δυνατότητα τη επαλήθευση τη κατάσταση πριν αυτή δημοσιευτεί. Και όλα αυτά πρέπει να παίρνουν χρόνο βεβαίω. Για να έχουμε λοιπόν ρεαλιστικέ προθεσμίε για την ανακοίνωση, για την κοινοποίηση τη κατάσταση, δύο δυνατότητε βλέπω ρεαλιστικέ. Πρώτον, να ζητούμε από την εταιρεία πριν από κάθε απογείωση να αποστέλλεται η κατάσταση επιβατών στην έδρα τη. Είναι δύσκολο μεν και ξέρω ότι δεν είναι όλε οι υπηρεσίε σύμφωνε, αλλά αυτό επιτρέπει τουλάχιστον σε ατυχήματο μέσα σε μία ώρα από το ατύχημα να επαληθεύει τον ε, τα ονόματα και τον αριθμό των μελών του, πληρωμά, πληρώματος η εταιρεία, χωρίς προβλήματα. Επίσης, όταν υπάρχουν συστήματα πρόορης ε, ειδοποίησης ή έγκαιρης προειδοποίησης για τους επιβάτες, μπορούμε τα στοιχεία αυτά να τα έχουμε διαθέσει μέσα σε 30 λεπτά. Γι' αυτά λοιπόν μπορούμε να συντονίσουμε το χρόνο, ενώ για τι άλλε πτήσει όπου δεν υπάρχει κατάσταση και δυνατότητα, μπορούμε να το παρατείνουμε στι δύο ώρε. Ένα άλλο ζήτημα είναι επίση πώ θα ενημερώνουμε του οικείου των θυμάτων. Ξέρετε ότι όταν συμβαίνει ένα αεροπορικό ατύχημα, χιλιάδε τηλεφωνήματα φτάνουν στα τηλεφωνικά κέντρα των αεροπορικών εταιριών. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ταυτότητα των θυμάτων, μάλιστα οι διαδικασίε ταυτοποίηση των θυμάτων είναι επώδυνε και πολύ επώδυνε για του οικείου. Θα πρότεινα λοιπόν, όπω γίνεται στι ΗΠΑ, να ζητούμε από τον επιβάτη κατά την κράτηση της πτήσης του να ορίζει κάποιον ε, υπεύθυνο να λάβει τη σχετική ενημέρωση. Πρόσωπο δηλαδή επαφή, κάποιο πρόσωπο επικοινωνία και βέβαια θα πρέπει να συζητήσουμε με τι αεροπορικέ εταιρείε το πώ θα γίνει αυτό στην πράξη, πώς θα εξασφαλιστεί αυτό στην πράξη, ταυτόχρονα με τον απόλυτο σεβασμό της, ε, των προσωπικών δεδομένων. Και εγώ θα ήθελα να έχουμε και ως δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των οικογενών για την διαξαγωγή και την εξέλιξη των ερευνών. Δεν ε, θεωρώ παραδεκτό να ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα αποτέλεσματα μιας έρευνας. Πρέπει να έχουν προνομιακή μεταχείριση, δηλαδή ε, πριν από όλου να ενημερώνονται και πάνω από όλο να λαμβάνουν και την προσωρινή αλλά και την τελική έκθεση διερεύνησης πριν από την δημοσιοποίηση και αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω των ενώσεων ή ομοσπονδιών οικογενειών ε, και οικείων θυμάτων. Ε, και κλείνω επίσης λέγοντας ότι στην παράγραφο 23, παράγραφος 1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ένα σχέδιο υποστήριξη των θυμάτων ε, της αεροπορικών ατυχημάτων και των οικείων τους, των οικογενειών τους, σε εθνικό επίπεδο. Πριν όμως η αεροπορική εταιρεία είναι ο πρώτος συνομιλητή, θα έλεγα, σε περίπτωση ατυχήματο. Θα πρέπει λοιπόν να πετούν τα κράτη-μέλη οι εταιρείε οι οποίε έχουν έδρα στα κράτη-μέλη του να έχουν και αυτέ αναπτύξει κάποιο σχέδιο κρίση, στο οποίο να περιλαμβάνεται και η ψυχολογική υποστήριξη. Επίση, η έρευνα ασφάλεια θα πρέπει να ορίζει και κάποιον ε, που θα αποτελεί το σημείο ή το άτομο επαφή για τι οικογένειε των θυμάτων. Εδώ το είδαμε αυτό ήδη και με το Ρίο και με το Γεμένια στη Γαλλία, με τηλεφωνική γραμμή ε, διαθέσιμη σε 24 ώρη βάση για, όλα τα, για όλες τις οικογένειες των θυμάτων και το ίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη δυνατότητα που δίνεται εκεί να ε, έρθουν ανα πάσα στιγμή, το χρειάζονται, οι οικογένειες των θυμάτων σε επαφή με τον αρμόδιο. Αυτό έχει βοηθήσει πολύ τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Και ταυτόχρονα μπορεί να υπάρξει καλύτερο τονισμός των πληροφοριών, από τα κράτη-μέλη και ναι, δίδεται και η ενημέρωση για τις διαδικασίες που αναπτύσσονται στη συνέχεια. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα πιστεύω και τις οικογένειες των θυμάτων που αισθάνονται χαμένες και σε αμηχανία ενώπιον των τόσων μεγάλων διαδικαστικών ε, δυσκολιών που ακολουθούν το μεγάλο τραύμα της απώλειας ενός αγαπημένου του προσώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και περιμένω τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας you, Mrs. κύριος Γκρός, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω στα γαλλικά. Έτσι θα με καταλάβει κατευθείαν η συνάδελφος. Συγχαρητήρια, είναι ιδιαίτερα τεχνική, αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητη η έκθεσή της. Για τα δίκτυα Δεν πιστεύω ότι αν όλη, όλη αυτή την προβληματική για την ε, συνοδευτική διαδικασία των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και την όλη ερευνητική διαδικασία. Δεν θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί αν τα επανεθνικοποιήσουμε όλα αυτά. Τώρα, για τους επιβάτες σίγουρα χρειάζεται ταχύτητα στην πληροφόρηση, αλλά χρειάζεται και αξιοπιστία. Δηλαδή η ταχύτητα δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της αξιοπιστίας. Θα πρέπει να υπάρχει μία εγγύηση μυστικότητας προς τα έξω, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνεται και όλη η πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. Τώρα, η ασφάλεια και η ανάλυση της ασφάλειας έχει προτεραιότητα, φτάνει να μην εμποδίζει την όλη δικαστική διαδικασία στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν για να μπορεί η δικαιοσύνη να δέχεται, να κάνει αποδεκτά ορισμένα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια, δεν θα πρέπει η ασφάλεια αυτή να προχωράει πέρα των νομίμων ορίων. Δεν θα πρέπει δηλαδή η ασφάλεια να παρακολεί τη δικαιοσύνη. Αυτά είχα να πω. Ο κύριος Αλχαντραούι, ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Ντεβεϊράκ για την προσέγγιση της αυτή και για το καλό της έργο. Πράγματι το σημείωμά της είναι εξαιρετικό. Κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πρώτα η συζήτηση για το δίκτυο εκεί. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, οπωσδήποτε δεν πρέπει να κάνουμε κανένα ένα βήμα προς τα πίσω και η πολιτική ερευνών να επανεθνικοποιηθεί. Νομίζω πως ε, το δίκτυο θα μπορούσε να είναι ένα ενδιάμεσο βήμα για ένα ευρωπαϊκό γραφείο, αλλά ας προσπαθήσουμε τώρα να μείνουμε σε αυτό το οποίο έχουμε για να ενισχύσουμε την δυνατότητα ερευνών και συμφωνώ πως πρέπει πράγματι να ορίσουμε καλά τον ρόλο και τα καθήκοντα του δικτύου. Νομίζω μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Δεύτερον, ΕΑΣΑ. Λέτε σύμβουλος, εντάξει. Νομίζω πως ε, πρέπει να ορίσουμε πάρα πολύ καλά πώς θα εμπλακεί κατά την διάρκεια της έρευνας και με τα δεδομένα της έρευνας και αν θα πρέπει να ενημερώνετε μονίμως. Γιατί βεβαίως μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από την έρευνα των ατυχημάτων που μπορεί να είναι σημαντικά όσον αφορά τα καθηκόντα πιστοποίησης της ΕΑΣΑ. Και είναι σημαντικό αυτό. Με τα δικαιώματα επιβατών. Η πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική στα μέλη των οικογενειών. Πράγματι, ε, όταν γίνεται κάτι πρέπει να το σκεφτούμε. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν τα άτομα τα οποία πρέπει να έρχονται σε επαφή όταν θα γίνονται οι ανακοινώσει. Ε, νομίζω πρέπει να το δούμε αυτό. Επίσης ο κατάλογος των υπηρετών πρέπει να δημοσιοποιείται το συντομότερο δυνατόν. Συμφωνώ και με ένα σχέδιο κρίσης για κάθε εταιρεία είναι εξαίρετο και να υπάρχει ένας μόνιμος για να είναι σημείο επαφής ανά εταιρεία. Εξαιρετική ιδέα. Τέλος, κάτι το οποίο σχετίζεται με την στατιστική, με τα στατιστικά ηχεία και τα σχετικά έγγραφα. Νομίζω πως εδώ πέρα πρέπει να ζητήσουμε να είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στατιστικά δεδομένα, να αναλυθούν, να ερμηνευθούν Οπότε σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη ε, να δουν τι θα γίνει με την υπάρχουσα βάση δεδομένων, ε, με την εισαγωγή δεδομένων και αυτή να γίνεται με τον ίδιο τρόπο παντού. Νομίζω έτσι θα, δώσουμε μια λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Ντεβεϊράκ για την έκθεση. Ε, πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που απαιτείται όμως γιατί βεβαίως μιλάμε για θανάτους σε αυτές τις περιπτώσεις και πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε. Ο κύριος Κατσίνος και ο δυσηγητής ε, δυστυχώς είναι απόν και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αιτίες αυτών των ατυχημάτων και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό να δούμε πώς θα μπορέσουν να αποφευχθούν στο μέλλον και νομίζω πως είναι αναγκαίο ακριβώς όπως το είπε και ο Ματιά να μην ξαναγυρνάμε σε κάποια επανεθνικοποίηση. Έχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα το τι θα γίνει με την ρύθμιση αυτών των θεμάτων και πρέπει να είναι αυτό προς το συμφέρον των ε, επιβατών που βεβαίως έχουν δικαίωμα να δουν μια βελτίωση εδώ πέρα. Επίσης αναφέρθηκε ο ρόλος της ΕΑΣΑ, πράγματι πρέπει να ξεκαθαριθεί, δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση συμφερόντων μεταξύ του τι κάνουμε εμείς τώρα ως δημιουργία δικτύου και την αρχική εργασία της ΕΑΣΑ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός, αλλά νομίζω ότι, όπως είπαν και οι προλύσαντες, πρέπει να συμπεριληφθεί η ΕΑΣΑ εδώ πέρα στις εργασίες και τέλος... Και εδώ πέρα νομίζω συμφωνώ με τον εισηγητή. Υπάρχουν κάποια ευαίσθητα δεδομένα με την εισηγήτρια που πρέπει να είναι κάπως ε, κρυπτογραφημένα. Δεν πρέπει να δίδονται γενικώ μόνο ίσως στη δικαιοσύνη, αλλά η προστασία των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τι θα δίδεται στη δημοσιότητα ε, όταν ε, ερευνούμε ένα στοίχημα ή δυσύχημα και τι όχι. Ευχαριστώ κύριο Ζένκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, εισηγήτρια για τις ε, πολύ χρήσιμε πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Το σχέδιο εδώ πέρα που ελπίζουμε να υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο έχει τους εξής στόχους. Να ερευνούμε τα ατυχήματα τα αεροπορικά ατυχήματα ε, με σκοπό βεβαίως να δλούνται διδάγματα για το μέλλον. Οπότε θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα θεμελιώδες ζήτημα γιατί σήμερα τα ερευνούν τα κράτη-μέλη τα ατυχήματα έχουν τις δικές τους υπηρεσίες ε, που ασχολούνται με την διερεύνηση ατυχημάτων και όταν αυτές οι επιτροπές ε, δεν ε, μοιράζονται τις ε, πληροφορίες, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Μόνο 50% των κρατών μελών έχουν ένα κεντρικό αρχείο. Αυτό είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Γνωρίζουμε πόσα ατυχήματα επαναλαμβάνονται και υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι αεροπλάνων, καμιά ε, δεκαριά. Οπότε πλέον ο εξοπλισμός είναι όλο και πιο τυποποιημένος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εξαναγκάσουμε τις υπηρεσίες των κρατών μελών να μοιραστούν τις πληροφορίες που έχουν. Γιατί όπως σας είπα έχουμε πληροφορίες μόνο από το 5% των ατυχημάτων. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, τα θύματα. Βεβαίω, είναι αποτελέσματα των ατυχημάτων, συχνά μεγάλων ατυχημάτων και αυτό το οποίο προτείνω εγώ είναι το χρονικό όριο ειδοποίηση των οικογενών να είναι το συντομότερο δυνατόν. Δεν συμφωνούμε με την δυνατότητα διαφορετικών ε, προθεσμιών σε διαφορετικές περιπτώσεις. Το σύστημα που έχουμε σήμερα περί ειδοποίησης των οικογενειών δεν είναι καλό γιατί ε, λαμβάνει υπόψη είναι τις νομικές πτυχές αλλά όχι τον ανθρώπινο παράγοντα. Επαφές με ψυχολόγους, δηλαδή γιατρούς και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Ναι, η σκιώδηση συγγήτρια η κυρία Λίχτενμπέργκερ δεν είναι εδώ, αλλά και εκείνη σας ευχαριστεί για την έκθεση, για τη συνεργασία. Πήγαν όλα καλά. Θέλω να αναφέρω δύο σημαντικά για εμάς ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το σημείο 5. Το υποστηρίζουμε πάρα πολύ. Γιατί τα θύματα δεν πρέπει μόνο να ενημερώνονται άμεσα για να μην έχουν αβεβαιότητες, αλλά και οι πληροφορίε περί της αποζημίωσης δεν μπορεί να τραβάει χρόνια αυτή η υπόθεση ε, καθώς απογοητεύονται με τα, τα θύματα. Πρέπει να υπάρχει μία προθεσμία για την καταβολή των αποζημιώσεων ή να γίνεται αμέσως. Ε, εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορεί να είναι ε, η πιθανώς δηλαδή νομική αντιπαράθεση να είναι εις βάρος των θυμάτων. Κατόπιν 5β ε, λέτε πως δίνονται πληροφορίες μόνο σε περίπτωση ατυχήματος όπου πρέπει κάποιος να ειδοποιηθεί και πρέπει να είναι άτομο έμπιστο κάποιος οικείος. Αλλά το υποστηρίζουμε, αλλά τα δεδομένα αυτά πρέπει να μην μεταδίδονται κάπου παραπέρα βεβαίως. Είδαμε και το πρόβλημα της συμφωνίας SWIFT, όπου όλες οι πληροφορίες μετά μεταδίδονται σε άλλους και δεν ξέρουμε σε ποιον πάνε. Ε, και μιλάμε για εμπιστευτικές ε, πληροφορίε. Εμπιστευτικές είναι και εμπιστευτικέ πρέπει να παραμείνουν και ανάλογος να είναι ο χειρισμός τους. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καταρχάς θα να ευχαριστώ την κυρία Τεβεγάκη που οργάνωσε την προκατακτική συνεδρίαση στην οποία είχαμε την ευκαιρία σύντομα να συζητήσουμε τις προθέσεις της. Χαίρομαι για την ανταλλαγή απόψεων και ε, για τις ε, τοποθετήσεις κυρίας Τεβεγιάκ και θα ήθελα ειδικά, ε, και έχω επί 25 χρόνια ασχοληθεί με την ε, ε, αεροπορική βιομηχανία από πλευρά κατά την επαγγελματική πεζοδρομία και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να συλληπιθώ τους εκπροσώπους των οικογενειών θυμάτων για τον πόνο τους. Αλλά θα ήθελα να πω ότι ό,τι έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια το έχουμε κάνει λόγω της βούλησης πολιτικής, λόγω της βούλησης για ανεξάρτητες διαρευνήσεις και λόγω της και χάρη στην πρόθεση να εξετάσουμε ε, μέχρι τέλους κάθε μηχανικό ε, σφάλμα ή ε, κάθε ανθρώπινο λάθος. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την, στην άκρη τη διερεύνηση Ενό ατυχήματο. Έτσι λοιπόν, ναι, μπορούμε να μιλούμε για δίκτυα, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει αυτό το δίκτυο να, υφί, να στηρίζεται πάνω στις υφιστάμενες ε, και εθελοντικές ε, συνεργασίες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιβάλλουμε νέα γραφειοκρατικά συστήματα τα οποία θα ε, επηρεάσουν σημαντικά την ελαφρά και ανεξάρτητη γραφειοκρατική δομή που έχουμε. Επίσης για τα άρθρα 8 και 9 η ομάδα εργασία από τα κράτη-μέλη, από του εμπειρογνώμονε των κρατών μελών, από ό,τι ξέρω, Πρόεδρε, έχει ήδη συνέλθει μετά τη σύνταξη του σχετικού κανονισμού, γιατί ήδη υπήρχαν κάποιε ανησυχίε και θέλαν να τα συζητήσουν. Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν, γιατί δεν πρόκειται να τα συζητήσουμε μέχρι τι 28 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθο, να δούμε κάποιε ιδέε για τι προτάσει αναδιατύπωση των άρθρων 8 και 9 που έχουν προτείνει οι πραγματογνώμονε. Αυτά τα άρθρα που μα απασχολούν εδώ. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να αποφύγουμε συγκρούσεις ε, συμφερόντων μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών Διερεύνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και της Επιτροπής. Ε, να ξέρει ο καθένας που εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή τη δουλειά θα κάνει χωρίς να θέλω να ε, επικρίνω κανέναν. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και σε αυτό που είπε η Κριστίν Βεράκ, νομίζω συμφωνούμε οι περισσότεροι. Ο ρόλος, ο συμβουλευτικός πάνω απ' όλα είναι σημαντικός Και καλό θα ήταν ίσως στο τέλος ε, η λέξη advisor να γραφτεί με όμικρον και όχι με air. Με συγχωρείτε που είμαι τόσο ψηλολόγος σε αυτά. Ε, νομίζω όμω ότι μπορούμε να παραπέμψουμε και στο άρθρο 13 τη Σύμβαση του Σικάγου, γιατί ό,τι και να λέμε, Πρόεδρε, εδώ έχουμε να κάνουμε με διεθνεί μεταφορέ, μιλούμε με για διεθνεί κανόνε και διατάξει, και άρα πρέπει η διατύπωσή μα να είναι απόλυτα ακριβή. Όταν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε διατύπωση, να υπάρχει η δυνατότητα τη επακριβού μεταφορά στο ε, δίκαιο τη εφαρμογή των νομοθεσιών, χωρί προβλήματα σχέση με τι διεθνεί ε, διατάξει και συμβάσει. Ξαναγύρισα λοιπόν στο σύμβουλο, advisor, που είναι η σωστή λέξη, ε, για δε το ρόλο ή την ερμηνεία του Συμβούλου. Ε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ της ε, ΕΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Οργανισμού Διερεύνησης των Εθνικών Αρχών και ιστορικοί λόγοι την έχουν υπαγορεύσει. Έτσι λοιπόν όταν μιλούμε για συμβουλευτικό ρόλο νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη επιλογή γιατί δεν μπορεί η ΆΤΑ να κάνει την ίδια δουλειά με τις υπηρεσίες διερεύνησης όπως σωστά είπατε και όπως άλλωστε αναφέρεται στην παράγραφο 2. Για το άρθρο 12. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και αντίστοιχα δικαιώματος προς την πρόσβαση στο μαύρο κουτί και τις καταστάσεις των επιβατών. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία από τα μαύρα κουτιά ε, και για αυτό το λόγο και δεν πηγαίνουν ούτε καν στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας. Υπάρχουν σαφείς λόγοι για τους οποίους οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί διαρεύνησης δεν κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά. Ε, στο σημείο 16 τώρα, ο αριθμός των μελών του πληρώματος έχει πολύ μεγάλη σημασία ασφαλώς, ε, αλλά δεν αφορά στοιχεία ε, που ανήκουν αποκλειστικά στα, στα μέλη του πληρώματος, δεν μπορούν δηλαδή να έχουν την αποκλειστικότητα στη χρήση ε, αυτή, είτε οι εταιρείε είτε κανείς άλλος, μόνο οι ε, οργανισμοί διερεύνησης. Και επίσης τα στοιχεία, τα σχετικά με τους επιβάτες, γιατί μιλούμε για κατάσταση επιβατών και όχι κατάλογο, ε, παραπάνω στοιχεία σχετικά με, τον, ε, με το άτομο επικοινωνίας ή επαφής, ίσως θα πρέπει να τα δούμε κάπως πιο προσεκτικά. Και ενώ θα πρέπει να πούμε σε προς λεπτομέρειες αργότερα, δεν θέλω να αφαιρθώ πρώτα στη δικαστική εξουσία, επειδή έχουμε διαφορετικές ε, δικαστικές παραδόσεις στις χώρες μας. Βλέπουμε ορισμένα πράγματα διαφορετικά εμείς. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και να κρίνουμε ίσω με διαφορετικό μάτι σε σχέση με την εμπλοκή του δικαστικού, τη δικαστική εξουσία. Στο κείμενο λοιπόν μπορεί ο ρόλος ε, ή μάλλον οι δηλώσεις των ε, ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας ή η δυνατότητα αυτές οι συνεντεύξεις και οι δηλώσεις τους να χρησιμοποιηθούν εις βάρος τους σε ε, δικαστικές διαδικασίες. Ο κίνδυνος της ενοχοποίησης ε, μέσω αυτών των δηλώσεων των ίδιων των ελεκτών, δηλαδή να βρεθούν οι ίδιοι υπόλογοι επειδή έκαναν κάποιε δηλώσει. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά γιατί έχουν μεγάλη σημασία ανάλογα με το νομικό σύστημα στο οποίο υπαγόμαστε. Και επίση θα ήθελα να επισημάνω στην εισηγήτρια. Ναι, πρόεδρε, τελειώνω σιγά σιγά. Έχουμε... Έχω και σκιώδη και συντονιστή, άρα μιλώ εκ μέρου δύο παραγόντων. Όχι, Πρόεδρε, εμεί από την ομάδα μου πάντα λογικά διαχειριζόμαστε το χρόνο μα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα κλείνοντα να πω ότι η συζήτηση σχετική με τη βάση των δεδομένων και τι σχετικέ πληροφορίε. Νομίζω ότι πρέπει στα όσα θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε σε επίπεδο της Επιτροπής μας, Πρόεδρε, και το έχετε δει και εσείς, Πρόεδρε, νομίζω ότι έχετε τη σχετική ενημέρωση. Ένα σύστημα έχει εισαχθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Είχαμε ζητήσει δηλαδή να υπάρχει το σύστημα της εθελοντικής ενημέρωσης που έχει λειτουργήσει στο Ρωμανό Βασίλειο αποτελεσματικά εδώ και 20 χρόνια και που έχει αποδείξει την αξία του και την αποτελεσματικότητά του. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όταν ε, κλείσει αυτή η υπόθεση, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη σε αυτό το πεδίο. Και κλείνοντας με αυτό, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Τεβεγάκ και να πω ότι πιστεύω πως θα έχουμε επικοδομητικό διάλογο και ότι θα καταλήξουμε, πιστεύω, γρήγορα σε καλά αποτελέσματα. Αλλά, όπως είπα, περιμένω κάποιε διευκρινήσει και από την Επιτροπή για την διατύπωση που έχει επιλέξει ορισμένα σημεία. Ευχαριστώ, κύριο Higgins. Thank you very much, Mr. President. I... Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα βεβαίω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους ε, Πάει να μπαίνει εδώ πέρα που έχουν τόσο πολύ υποφέρει από το θάνατο των οικείων του και βεβαίω ο στόχο μα εδώ πέρα είναι να φροντίσουμε ότι θα είναι το δυνατόν πιο λεπτομερείς οι έρευνε για να οδηγηθούμε σε πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά που ήδη ακούστηκαν. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να έχουμε ανεξάρτητε έρευνε και να συμβαστεί και ο δικαστικό ε, και ο ρόλο ασφάλεια. Και βεβαίως όσον αφορά την απελευθέρωση πληροφοριών, το ποιος είναι δηλαδή, ποιος επιβαίνει σε ένα αεροσκάφος όταν αυτό πέφτει, να δίνεται προτεραιότητα στους συγγενείς και όχι στα ΜΜΕ. Αυτοί πρέπει να ενημερώνονται πρώτοι. Υπάρχουν δύο πτυχές εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα η έρευνα και δεύτερον η πρόληψη. Να πω πως πριν από λίγε εβδομάδες είχαμε μία ομάδα πιλότων εδώ απ' έξω που έδιναν μοίραζαν φυλάδια για τις ανησυχίες τους για την ε, μείωση στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών όσον αφορά τις ώρες εργασίας τους. Εγώ είμαι υπέρ του ανταγωνισμού και της μείωσης του κόστους, αλλά οι πιλότοι φύσανται τεράστια πίεση. Παραδείγματος χάρη μια αεροπορική γραμμή της χώρας μου, της Ιρλανδίας, έχει χώρο μεταξύ πτήσεων 20 λεπτά είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους και ανησυχία στον, ε, για την ασφάλεια. Και μάλιστα συμπτωματικά την τελευταία, στην τελευταία μου πτήση καθόμουν ε, δίπλα σε έναν πιλότο της Air Lingus που ήταν εδώ στη διάσκεψη και σημαντικό κομμάτι της διάσκεψης ήταν η πίεση που ασκείται στους πιλότους. Έχουν πλέον πολύ περισσότερες ώρες που πρέπει να δουλεύουν, είναι εξαντλημένοι και μιλάμε για μεγάλο κομμάτι της αεροπορικής ασφάλειας. Εμείς μιλούσαμε για την ασφάλεια από κακόβουλες πράξεις, ανιχνευτές σώματος κτλ. Επίσης ήμασταν πάρα πολύ αυστηροί στην ασφάλεια από οδικά ατυχήματα, αλλά ασφάλεια από ατυχήματα σε αεροπορικές μεταφορές όσον αφορά την πίεση που ασκείται στους πιλότους και το ότι έχει μειωθεί και εκπαίδευση. Είναι κάτι το σημαντικό για να μειωθούν ε, τα ατυχήματα και τα θύματα. Αυτά και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άλβαρες. Gracias, Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, συμμερίζομαι. Και εγώ το πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση. Είναι πολύ ασφαλής οι αερομεταφορές. Όμως από καιρού εις καιρών γίνονται δυστυχήματα και θέλουμε εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε όταν γίνεται ένα δυστύχημα να διελευκάνουμε τις αιτίες. Τώρα, για τα μέτρα που μπορούν να, απαλει... να αμβλύνουν τον πόνο των συγγενών. Εγώ ξέρω ε, κάποιον ε, που είχε συγγενείς στο δυστύχημα της Σπανέρ ε, και ξέρω τι μπορεί να τραβήξει κανείς όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί απάντηση. Εγώ λοιπόν Συμφωνώ με την εισηγήτρια να έχουμε τον κατάλογο των επιβατών πριν από την απογείωση του αεροπλάνου. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ, σύμφωνα με τη σύμβαση του Σικάγου, ότι δύσκολα μπορεί να έχει η εταιρεία τον κατάλογο των επιβατών πριν από την απογείωση. Η μία ώρα για αυτούς που περιμένουν νέα είναι ένας αιώνας και οι δύο ώρες είναι αιωνιότητα. Μου φαίνεται λοιπόν αδιανόητο να μην ξέρουν οι εταιρείε ποιος ταξιδεύει στα αεροπλάνα τους. Επίσης, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και για το τι εμπορεύματα κουβαλάει αυτό το αεροπλάνο. Πολλές φορές μπορεί να κουβαλάει επικίνδυνα φορτία, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Και επίσης θα πρέπει να βρούμε μία λύση που να μην αντιπαραθέτει την έρευνα για τις αιτίες του δυστυχήματος με την δικαστική έρευνα. Ευχαριστώ κύριος Φαντάλεν, ο Αντιπρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα περιοριστώ σε λίγα πραγματάκια προς την κυρία Βεϊράκη, γιατί ο χρόνος πιέζει πρώτα απ' όλα. Στην παραγραφό 4 λέτε πως φαντάζεστε πως Ό,τι προκύπτει από την ανάλυση πρέπει να πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Εγώ στο παρελθόν ε, έχω λάβει μέρος σε πολλές διερευνήσεις ατυχημάτων και η αίσθησή μου είναι πως ε, ήταν άμεσα εκεί πέρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ζητήσει δεδομένα. Αλλά σημαντικό είναι να υπάρχει κάποια ανεξαρτησία στην ε, έρευνα και θα πρέπει να κάνει πρώτα απ' όλα τα καθήκοντά του αυτός ο οποίος κάνει διερεύνηση και να μην ε, είναι αμέσως επάνω του το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οπότε έχουμε εμεί έναν εξάρτητο Συμβούλιο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων στην Ολλανδία και πηγαίνουν ε, τα στοιχεία στη δικαιοσύνη μόνο όταν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη, τρομοκρατία, ε, θάνατος ή ομοιρία και δεν πηγαίνουν όλα τα στοιχεία κάθε ανάλυσης. Δεύτερον, η υποχρέωση ενημέρωσης, κάποια πράγματα έχετε και εδώ πέρα, ναι. Επαφίεται στην δικαιοσύνη ο τρόπος ε, επέμβασης. Δεν ξέρω αν είναι επιθυμητή αυτή η κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια για την υποχρέωση ενημέρωσης που θα έπαιζαν ένα ρόλο όσον αφορά την ενημέρωση. Θα ήθελα να περιοριστεί λίγο εδώ πέρα ο ρόλος δικαιοσύνης για να είμαστε και σύμφωνοι με την συνθήκη του Σικάγου. Επίσης μίλησαν κάποιοι συνάλφοι για ένα ευρωπαϊκό γραφείο. Δεν είμαι σίγουρος, εκτός εάν διαλέξουμε έναν τρόπο ο οποίος θα διασφαλίζει Πλήρω την ανεξαρτησία. Γιατί βλέπω πως κάποια κράτη-μέλη από τη μία έχουν μία αστυνομία αεροπορίας, οπότε επεμβαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, και φοβάμαι πως ε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει η απαραίτητη ανεξαρτησία για να μπορέσουμε και να διδαχτούμε από αυτά τα περιστατικά τα ατυχήματα. Σας ευχαριστώ η κυρία Γιάλα Σέντερ presidentes, y felicitar Να συγχαρώ την εισηγήτρια για τον τόσο προσεκτικό τρόπο που προετοίμασε την έκθεση. Τώρα, για την ΕΟΑΑ και την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Εμείς βλέποντας το τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τα διάφορα δυστυχήματα όπου έχουμε την έρευνα για την αιτία του δυστυχήματος και τη δικαστική έρευνα βλέπουμε πολλές φορές λοιπόν να υπάρχει αδυναμία πραγματογνωμοσύνης και μεταβίβασής της στα δικαστήρια και το γεγονός ότι η έρευνα δεν κοινοποιείται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, ούτω ώστε να μπορεί κανείς να προσφεύγει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας να ζητάει μία εξπερτής. Και θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα του όταν ζητούνται διερευνητικά στοιχεία από τη δικαιοσύνη, ορισμένα να δίνονται και ε, ορισμένα όχι, άλλες φορές ναι και άλλες φορές όχι. Και αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δυστυχήματα, Για τα δυστυχήματα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα για την αναγνώριση των θυμάτων. Εμείς στην Ισπανία έχουμε ένα σύστημα, ας πούμε στο κινητό, να, υπάρχει και το όνομα του ιδιοκτήτη, πράγμα το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για να γίνεται η ταυτοποίηση όταν έχουμε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα αεροπορικά δυστυχήματα. Υπάρχει πάντα βέβαια το πρόβλημα σε ποιον πρέπει κανείς να, να ανακοινώσει έναν θάνατο, ε, με ποιον τρόπο κλπ. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των αεροδρομίων. Και πρέπει να υπάρχει και η πρόληψη. Δηλαδή, να γίνεται η διερεύνηση και η κοινοποίηση αυτής της διερεύνησης ως κομμάτι της πρόληψης. Κύριε ε, σύντομα μόνο για τον κατάλογο των επιβατών ή την κατάσταση. Δεν βλέπω γιατί η Πρόεδρε δεν μπορεί να έχει ένα διεξοδικό, μια διεξοδική κατάσταση επιβατών μια αεροπορική εταιρεία πριν την απογείωση του αεροσκάφου. Κανένα λόγο δεν βλέπω. Έχουμε τις πληροφορίες. Υπάρχει το φορτίο στην κατάσταση του αεροσκάφου, το λεγόμενο μανιφέστο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να συζητάμε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι το κάνουμε αυτό. Αυτές τι πληροφορίες θα τι κάνουμε εάν χρειαστεί ομιγέννητο. Αυτό είναι μόνο. Αλλά δεν μπορείτε να μας λέτε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αυτέ οι καταστάσεις. Πρόεδρος. Εντάξει. Σημειώνουμε την παρατήρησή σας. Πριν ε, να ζητήσω από τον κύριο Σέιμπομ με την Επιτροπή να μας ε, κάνει δικέ του παρατηρήσει, σα κάνω και εγώ μερικέ παρατηρήσει αν μου επιτρέπετε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό και με την κυρία Φώστερ και με τον κύριο Φαντάλεν ως προς το ρόλο της ΕΑΣΑ. Ανησυχώ δηλαδή ότι η ΕΑΣΑ, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό, δηλαδή, μπορεί να, η ΕΟΑΑ, μπορεί να θεωρηθεί ως ισότιμος εταίρος σε μια τέτοια έρευνα που πρέπει να αποφύγουμε βέβαια. Δεν μπορεί η ρυθμιστική αρχή να είναι ταυτόχρονα και ερευνητική αρχή ή να συμπράττει με τις ερευνητικές αρχές. Έτσι λοιπόν, από την ΙΚΑΟ και από τη Σύμβαση του Σικάγου και το 13ο παράρτημα, είναι ξεκάθαρο ότι έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα η παρουσία ε, ενός του οργανισμού. Σε αυτό δεν έχω καμιά αντίρρηση. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν ήταν αμερικανικό αεροσκάφο, θα είχαμε και αμερικανική αρχή. Αν ήταν γαλλικό αεροσκάφο, πάλι θα είχαμε του εκπροσώπου τη γαλλική αρχή ω συμβουλευτική όμω παρουσία, μόνο με συμβουλευτικέ ε, αρμοδιότητες. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Άλλο πράγμα είναι η διερεύνηση ενό ατυχήματο και άλλο είναι η παρουσία και ο ρόλο τη ε, ρυθμιστικής αρχής. Γιατί μπορεί να έχει τελευταία ανάλυση και ίδιο συμφέρον η ρυθμιστική αρχή. Μπορεί κάποιο σφάλμα δικό της να έχει οδηγήσει στην, ε, στο ατύχημα στην πτώση του αεροσκάφου. Μπορεί γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν βέβαια και οι μαύρες λίστες ε, από την ΙΚΑΟ και τα λοιπά, όλα αυτά μπορεί να οφείλονται, ένα ατύχημα μπορεί να οφείλεται σε κάποια παράληψη ή πράξη της ρυθμιστικής αρχής και όχι στις εταιρείε. Επομένως δεν μπορούμε, και καλά κάνουμε η κυρία Βεϊάκ, Βεϊάκ, να μπερδεύουμε το ρόλο της ε, ε, ρυθμιστικής σε κυρια βειακ βειακ να μπερδευουμε το ρολο της ρυθμιστικης αρχης με το ρόλο μιας ερευνητικής αρχής. Μόνο συμβουλευτικά όπως είπα. Επίσης προς τον τόπο του ατυχήματος, γιατί πάντοτε βλέπουμε κατάπληξη. Και το είδαμε και με το τελευταίο συνδρομικό ατύχημα στο Βέλγιο. Έρχονται πάντα κάποιοι, 5 λεπτά ή 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μέσω μετά το ατύχημα, να πούνε Α, ξέρω εγώ για ποιο λόγο. Συνήθω αυτή εμφανίζεται στα ΜΜΕ, αλλά όπω και να έχει, πάντα κάποιο προσπαθεί να μα εξηγήσει του λόγου που οδήγησε σε ένα ατύχημα. Και εμεί που ξέρουμε πολύ καλά τι μεταφορέ, ξέρετε πόσο, πόσο σκληρά αγωνιζόμαστε να λέμε, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να μιλάτε για αιτίε ατυχήματο μέχρι ότου ετοιμαστεί η επίσημη έκθεση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι να την λέγουν «Α, εγώ ξέρω» και ε, να χαρακτηρίζουν τον τόπο του ατυχήματος ως τόπο εγκλήματος. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως έγκλημα παρά μόνο αν ξέρεις ότι είναι έγκλημα, ότι υπάρχει εγκληματική ε, πρόθεση ή δραστηριότητα. Είναι μια ε, τόπος τραγωδίας, αν θέλετε, τόπος ατυχήματος, αλλά δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τόπο εγκλήματος. Άρα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς, τι έχει οδηγήσει στο ατύχημα, εάν έχει να εμπλακεί η δικαιοσύνη και ποιος θα κληθεί να λογοδοτήσει. Τρίτον όμως με τη σειρά. Εάν τα μπερδέψουμε όλα αυτά και ανατρέψουμε τη σειρά, μπορεί κάποιοι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι μπορεί κάπως να γνωρίζουν τα πράγματα, μπορεί να ξέρουν τι έχει πάει στραφά, να τρομάξουν και να μην μιλήσουν ξεκάθαρα φοβούμενοι ότι μπορεί να ξεκινήσουν εις βάρος τους δικαστικές διαδικασίες, εις βάρος κάποιου συναδέλφου. Και εγώ δεν λησμονώ ποτέ τον ε, ελεγκτή ενέργειας κυκλοφορίας που δολοφόνησε ο πατέρας ενός θύματος ενός ε, ε, ρωσικού δυστυχήματος που είχε συγκρουστεί με ένα γερμανικό. Χωρίς να ξέρει αυτός ο άνθρωπος τι είχε συμβεί, πήγε και δολοφόνησε τον ελεγκτή αέρας κυκλοφορίας. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν αυτά να... Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτές τις υποθέσεις. Και ευχαριστώ την κυρία και είναι πολύ καλή έκθεση και πολύ καλές συζητήσεις. Ε, πάντως συμφωνώ και εγώ απολύτως με τα όσα υπόθηκαν εδώ για, από πολλούς συναδέλφους. Ιδιαίτερα πάντως η κυρία ε, Φώστερ και ο κύριος Φαντάλεν, πρέπει να το επισημάνω. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί όταν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Και πάνω απ' όλα να διαφυλάσσουμε την ανεξαρτησία και τις διευχωριστικέ γραμμές του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και των Ερευνητικών. Η κυρία Ντεβιγά, αλλά πρώτα η Επιτροπή. Με συγχωρείτε, Παρασύρθηκα. ο κύριος Σέιβα από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ την εισηγήτρια για μια πρώτη σημερινή συζήτηση. Νομίζω το έγγραφό της είναι όντως ε, πολύ επιτυχές και ανταποκρίνεται στα ίση παρατήρηση Επιτροπής, καλύπτει όλα τα ζητήματα, νομίζω ότι αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση. Επίσης θεωρώ ότι αυτή η πρώτη συζήτηση ήταν μια πολύ ειλικρινής παράθεση απόψεων. Και άρα αποτελεί ένα καλό ιονό για περαιτέρω ειλικρινής ανταλλαγής απόψεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στρα από 15 χρόνια, που είχαμε την πρώτη οδηγία για τη διερεύνηση των ατυχημάτων, καταθέτει προτάσει για περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματο αυτού και στηρίζεται πάνω σε δύο βασικέ γραμμέ, Πρόεδρε. Καταρχά, έχοντα αξιολογήσει την μέχρι τώρα εμπειρία μα, θετική μεν αλλά και όχι τόσο θετική εμπειρία, που κατά την άποψή μα σημαίνουν ότι χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, από τα 15-7 χρόνια εμπειρία που έχουμε, βλέπουμε ότι ήρθε η ώρα πλέον να στήσουμε από τα εθνικά νομοθετικά συστήματα να μας δώσουν απαντήσεις για το αν έχει βελτιωθεί η ασφάλεια των αέριων μεταφορών και αν υπάρχει δυνατότητα για αντίστοιχη βελτίωση και της διερεύνησης των ατυχημάτων. Δεν θα επισέλθω στι ενδιαφέρουσε κατά τα άλλα παρατηρήσεις που ακούστηκαν στη λεπτομερία τους. Απλώς θέλω να σημειώσω ότι χρειάζεται εξυγχρονισμό του συστήματος, αυτό το ομολογούν όλοι. Αυτό έχουμε προτείνει και εμείς. Η ουσιαστική μα στόχη είναι πρώτον η βελτίωση του ερευνητικού δυναμικού της δυνατότητας για την ερεύνηση ατυχημάτων στην Ευρώπη εν γέννη με την επιβέωση και την ενίσχυση ενός δικτύου των υφισταμένων αρχών ενός δικτύου που ήδη υπάρχει, αλλά που πιστεύουμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί ως προς το ρόλο του, περαιτέρω, και επίσης, Πρόεδρε, έχοντας υπόψη και την ε, ε, δυνατότητα για ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων σε αυτό το δίκτυο, για πιο καλή ανταλλαγή απόψεων, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και των ε, γνώσεων των ε, πραγματογνωμόνων. Έχουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη πολύ καλά αποτελέσματα, σε άλλα λιγότερε δυνατότητε, λιγότερα μέσα και πόρου και ίσω μπορούμε χάρη στο δίκτυο αυτό να βοηθήσουμε εκείνα τα κράτη που έχουν περισσότερε δυσκολίε για τη διερεύνηση. Δεύτερο, ένα σημείο το οποίο αρκετοί ε, βουλευτές της Επιτροπής σας επισήμαναν, στο παρελθόν και μέχρι σήμερα έχουμε δει αρκετέ φορέ συγκρούσει μεταξύ τη διερεύνηση του ίδιου του ατυχήματο, δηλαδή των αιτιών του ατυχήματο και τη ε, διαδικασία ανακριτική ή δικαστική που μερικέ φορέ χωρί ω κακή πρόθεση έχει παρεμποδιστεί λόγω αυτή τη ε, ανάμειξη των διαδικασιών και γι' αυτό χρειάζεται μια σαφή διαχωριστική γραμμή. Τρίτον, έχουμε ήδη και το έχουμε επισημάνει εξασφαλίσει μια καλή νομοθεσία στην Ευρώπη για την ασφάλεια. Έχουμε μια υπηρεσία ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό οργανισμό που ασχολείται με τα θέματα της ασφάλειας και ως εκ τούτου πιστεύω απαιτείται η σχέση μεταξύ του οργανισμού αυτού και των ερευνητικών ε, υπηρεσιών, των υπηρεσιών διερεύνησης, να διευκολυνθεί, να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία όπως είπαμε, ε, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, επισημαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ε, όταν ε, ο οργανισμός αναλαμβάνει ερευνητικό ρόλο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας είναι γνωστό και δεν περιορίζεται μόνο στα φαινόμενα των ατυχημάτων των αεροπορικών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν αντιμετωπίσει και συζητήσει εξωτικά και στις ΗΠΑ οι αρχές, όπως σε παραδείγματι ειδικότερα σε περίπτωση ατυχήματος, τι ακριβώς καλείται να διερευνήσει ο οργανισμός ο ρυθμιστικός και τι η υπηρεσία διερεύνηση. Σε πάση περιπτώσει όμως δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα ενός συμβουλευτικού ρόλου της ΕΟΑΑ ε Καταρχάς διότι έχει την εμπειρία ως ρυθμιστικός οργανισμός, έχει τις γνώσεις να βοηθήσει και να κατευθύνει σε πιο στοχευμένα αποτελέσματα τις έρευνες, αλλά ταυτόχρονα και γιατί μπορεί να ε, ε, εποφεληθεί από την ερευνητική αυτή διαδικασία για να αποτρέψει στο μέλλον την επανάληψη αντίστοιχου ατυχήματος για τους ίδιους λόγους. Άλλο ένα σημείο για την ε, ασφάλεια. Σε περίπτωση που επισημαίνεται μια σειρά πιθανών αιτιών ύστερα από ένα ατύχημα, μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις ασφάλειας πριν από την ε, εκκίνηση διαδικασίας για την αναθεώρηση της νομοθεσίας, πριν από την ε, τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό προτείνουμε να υπάρξει μία βάση δεδομένων για κάθε ενδιαφερόμενη αρχή που θα μπορούσε να χρήσιμη για αυτό το σκοπό. Και ένα τελευταίο σημείο στο οποίο αναφερθήκαμε ε, ήδη είναι τα δικαιώματα των οικείων των θυμάτων ως αεροπορικού ατυχήματος. Ε, συχνά με, το, με την ανακοίνωση ε, ενός ατυχήματος διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, δυσκολίες ε, και ταλαιπωρία των οικείων των ε, θυμάτων ή των επιβατών αν θέλετε. Πρέπει όμως να υπάρχει δυνατότητα και να έχουν μια κατάλληλη ενημέρωση για, τον, για τα ονόματα των επιβατών αλλά και να υπάρχει η κατάλληλη πρόσβαση των οικείων αυτών στις πληροφορίες σχετικές με το ατύχημα χωρίς βέβαια να προσβάλλει τη βασική αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτή είναι η πέντε βασική στόχη πρόεδρε νομίζω. και νομίζω ότι έχει εκφραστεί με την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων μια σαφή υποστήριξη στου στόχου μα. Λαμβανομένων φυσικά υπόψη και των εκάστοτε συμπληρωματικών ή επικριτικών παρατηρήσεων, τι οποίε θα λάβουμε με κάθε σοβαρότητα υπόψη. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει σε επίπεδο Συμβουλίου και υπό ε, Ισπανική Προεδρία με μια γενική προσέγγιση που έχει ξεκινήσει ήδη και θα δούμε εάν μπορούμε για το θέμα αυτό να προβλέψουμε ε, επικοινωνία και τα λέγει απόψε μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ε, στο ε, μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική και χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Χριστίν Βιγάκ, θέλεις να πεις δύο λόγια. Σύντομα υποθέτω. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να απαντήσω στον καθένα χωριστά. Ήσασταν πολλοί που μιλήσατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Αλχαδράουρη, η κυρία Μέσνερ ε, μίλησαν για τον οργανισμό. Πρέπει να ορίσουμε τις αρμοδιότητες. Αν ακούσουμε την κυρία Φόρστερ ή τον κύριο Βαντάλεν, φαίνεται ότι δεν είναι ασυζήτητο να προτείνουμε νέες υποδομές. Όλοι τοποθετηθήκατε για το πώς θα μπορούσε να μην είναι τόσο δυνηρή η αναγγελία στους ε, οικίους των επιβατών. Να δίνεται η λίστα των επιβατών όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και, αλλά όπως είπε και ο κύριος ε, Γκρός ε, θα πρέπει να δίνεται γρήγορα η λίστα, πρέπει να είναι όμως και αξιόπιστη. Τώρα ε, συνάδελφε εγώ σκέφτομαι, έχω, εγώ Εγώ κυρία Άλβαρες ε, τα ίδια πράγματα με εσάς σκέφτομαι αλλά ξέρετε πολλές φορές την τελευταία στιγμή υπάρχουν ε, επιβάτες ε, που αλλάζουν εισιτήρια, που αλλάζουν αεροπλάνα δύσκολα δηλαδή μπορεί κανείς να έχει μία αξιόπιστη λίστα αμέσως. Κύριε Κράμερ μιλήσατε για την εμπιστευτικότητα σχετικά με την επαφή. Ναι, γι' αυτό εγώ ορίζω ότι θα πρέπει ε, την εποπτεία να την έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προστασίας Δεδομένων. Με του Σάντοφ θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε το θέμα, αλλά βλέπω ότι σας ενδιαφέρει όλους. Που είμαι ανοιχτή λοιπόν, θα συζητήσουμε όλοι μεταξύ μας. Ευχαριστώ. 28 Απριλίου θα δούμε το σχέδιο έκθεσης. 4 Μαΐου προθεσμία για τροπολογίες. Ελπίζουμε πρώτη Ιουνίου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή και να πάει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Προθεσμία λοιπόν για τροπολογίες 4 Μαΐου, αλλά ελπίζουμε να γίνει άλλη μια συζήτηση στις 28 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο. Διεθνείς αεροπορικές συμφωνίες και διαδικασίες μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, δικό μου είναι αυτό το θέμα, μου το έδωσαν οι συντονιστές. Θα θυμάστε πως απαιτείται η συνένεση του Κοινοβουλίου πλέον με τη συνθήκη Λισαβόνας πριν συνάψει διεθνείς συμφωνίες ε, το Συμβούλιο με την κανονική δηλαδή νομοθετική διαδικασία, αυτό το οποίο λέγαμε παλαιά συναπόφαση, παλιά συναπόφαση. Οπότε πολλές από τις συμφωνίες που αφορούν την Επιτροπή μας, ειδικά οι αεροπορικές, απαιτούν και την συνένεση του Κοινοβουλίου και όχι μια απλή γνωμοδότηση όπως επί τις ε, διαδικασίες ε, της διαβούλευσης. Οπότε, εν ώψη του ενισχυμένου ρόλου μας, θεωρήσαμε πως καλό θα ήταν να κάνει μία παρουσίαση η Κομισιόν όσον αφορά τους στόχους της στη διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών. και το ποιε είναι πιθανόν να έρθουν για να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο του ερχόμενου μήνε. Ελπίζω να σωστά ανοιχθεί η εισαγωγή για τι μελλοντικέ συζητήσει. Οπότε, κατόπιν ετήματο των συντονιστών ζητήσαμε να έρθει η Κομισιόν να μας εξηγήσει την τρέχουσα κατάσταση. Ο κύριος είναι Μπουγκελβένε. ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας, που είναι προϊστάμενος της ε, αρμόδιας μονάδας. Έχετε τον λόγο. Merci, ε, Président. Ε, vous... Ευχαριστώ, Ότι κατά την προηγούμενη θητεία η Κομισιόν είχε παρουσιάσει μία ανακοίνωση για την πολιτική αεροπορία και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξή της στην Ένωση. Προσπαθώντας να έχουμε η ισότητα και αμοιβαιότητα στα θέματα ανταγωνισμού. Έχουμε λοιπόν δύο πυλώνες. Ένα ρυθμιστικό πυλώνα, ο οποίος θέλει να εγγυθεί τη νομική ασφάλεια των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών και αυτό μετά την απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2002, την απόφαση Open Sky. Υπάρχουν ε, γύρω στις ε, 80 και κάτι συμφωνίες, 40 έχουν επικυρωθεί και νομιμοποιηθεί μέσα από οριζόντιες συμφωνίες. Υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας τώρα που είναι ο οικονομικός πυλώνας και όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες με τους εταίρους μας ανοίγοντας ε, την αγορά των μεταφορών, με τους εταίρους κλειδιά και τις ε, γείτονες ε, χώρες ε, και, να με παιδίσεις στον τομέα αυτών. Να ξεπεράσουμε δηλαδή το κλασικό δικαίωμα στη διακίνηση και να έχουμε έναν ανοιχτό ουρανό Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα για τις συμφωνίες. Με τις Ηνωμένε Πολιτείε διαπραγματευόμαστε, έχουν προχωρήσει πολύ οι διαπραγματεύσεις ε, για να ανανεώσουμε τη συμφωνία που είχαμε από το 2007 και τον προηγούμενο Δεκέμβριο υπογράψαμε με τον Καναδά. Συνεχίζουμε διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία, με την, Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία Επίσης ζητήθηκε εντολή από την Κομισιόν για την Κίνα και την Ινδία. Αλλά ακόμη το Συμβούλιο δεν έδωσε αυτή την εντολή. Τώρα για τις ε, γείτονες χώρες θα πρέπει να μιλήσουμε για κοινό ενέργειο χώρο με τις ίδιες προδιαγραφές που θα βασίζεται στο δικό μας κεκτημένο. Έχουμε Μία παλιά συμφωνία με το Μαρόκο, το 2006 υπογράφτηκε. Έχουμε συμφωνία με τα Δυτικά Βαλκάνια και έχουμε και διαπραγματεύσεις που εκκρεμούν η Ορδανία, Λίβανο, Ισραήλ αλλά και την Ισία και Αλγερία σαν εγγύς μέλλον. Συζητάμε επίσης και με τη Γεωργία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η κατάσταση για τις αεροπορικές υπηρεσίες. Τώρα, παράλληλα, έχουμε ειδικέ συμφωνίες για την ενέργεια ασφάλεια. Συμφωνία λοιπόν του 2009 με τον Καναδά ή υπογραφή με τις Ηνωμένε Πολιτείε ή ακόμη υποδιαπραγμάτευση με τη Βραζιλία. Προς υπόμνηση, έχουμε μία συμφωνία συνεργασίας με την, οργάνωση, ε, τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας και μετά έχουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων ε, διαχείρισης εναερίου κυκλοφορίας από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Αυτά για να σας αναφέρω που βρισκόμαστε με τις διεθνείς αεροπορικές συμφωνίες. Αν θέλετε τώρα αναλυτικότερες πληροφορίες θα σας τις δώσουμε θα σας ετοιμάσουμε και θα σας ε, στείλουμε συντομότατα έναν αναλυτικότατο πίνακα που θα εξηγεί που βρισκόμαστε ακριβώς με τις διαπραγματεύσεις εκείνες που μάλλον με τις συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν καταλήξει ακόμα γιατί βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση και Για να μιλήσουμε τώρα για τους νέους όρους που απαιτεί η Λισαβόνα από το Κοινοβούλιο και αν η μνήμη μου είναι καλή για την παράγραφο 19 όπου τα μέλη της Επιτροπής σας θα πρέπει να ενημερώνονται για το πώς εκτιλίζονται οι διαπραγματεύσεις για τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον ε, Καναδά, διαφυλάσσοντας όμως και τη μυστικότητα αυτών των διαπραγματεύσεων. Η Συμφωνία Πλαίσιο του 2005 το έχει προλάβει αυτό το άρθρο το 218 τη δίνει στο Κοινοβούλιο τα μέσα άσκησης ενισχυμένης ε, νομοθετικής συνεργασίας. Επίσης, στις Ηνωμένε Πολιτείες θα συμμετέχει και ένα μέλος της Επιτροπής σας. Όλη αυτή η, εργασία, η διεργασία πληροφόρησης θέλει να αποδείξει ότι θέλουμε μία ισορροπία μεταξύ δηλαδή ρυθμιστικής ε, σύγκλησης και ανοίγματο των αγορών. Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Και το Κοινοβούλιο είχε δείξει αυτήν την